Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Χθες αργά το απόγευμα, Ε, είχαμε τη συνεδρίασή μα, ε, μοιράζονται αυτή τη στιγμή τα πρακτικά και θα θεωρηθεί ότι εγκρίθηκαν εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσει μέχρι το τέλος της συνεδρίασή μας. να σας ενημερώσω ότι η συνεδρίασή μας γίνεται με την παρουσία εκπροσώπων του Εμπορικού Επιμελητηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχαμε πρωινό γεύμα και ανταλλαγή απόψεων για, την, για τον γύρο της Ντόχα. Ελπίζω ότι θα υποφεληθούν από τη συνεδρίασή μας, να σας ενημερώσω. Σας παρακαλώ, λίγη ησυχία. Παρακαλώ προσέξτε με γιατί πρέπει να λάβουμε απόφαση. Να ξεκινήσουμε άτυπες ε, διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Κομισιόν για την επίτευξη συμφωνίας κατά την πρώτη ανάγνωση σχετικά με την ε, διμερή ε, εγγυητική ρήτρα της ε, Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωση Κορέα. Σύμφωνα με τις γενικές αρχές για τις διαδικασίες... Σας παρακαλώ, εδώ στα αριστερά, προσέξτε με. Έχει ξεκινήσει η συνεδρίαση. Οι συζητήσεις να γίνουν έξω από την αίθουσα. Σύμφωνα με τις γενικές αρχές μας για τις ε, επίσημες διαπραγματεύσεις ε, σε κανονικές νομοθετικές διαδικασίες που υιοθετήθηκαν από τους συντονιστές ε, στις 31 Στι 21 ε, Φεβρουαρίου φέτο ε, προτείνω να ε, λάβουμε την εξή απόφαση. Να ξεκινήσουμε επίσημε διαπραγματεύσει με την Κομισιόν και το Συμβούλιο για την επίτευξη συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση. Δεύτερον, να εγκρίνουμε την έκθεση, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την εντολή τη διαπραγματεύτική ομάδα και τρίτον, η διαπραγματευτική ομάδα να αποτελείται από εμένα, που θα προεδρεύω, τον εισηγητή μας, τον κύριο Φάλπερ και τους σχεδόν εισηγητές Λάγκε, Στέρντι, Φαέρα και Σόλτς. Αυτή είναι η επίσημη απόφαση που πρέπει να λάβουμε για να προχωρήσουμε με το θέμα αυτό. Υπάρχουν αντιρρήσεις ως προς την πρόταση αυτή. Όχι. Ωραία, θεωρώ ότι εγκρίθηκε. Να προχωρήσουμε λοιπόν στο σημείο 9. Εμπορικέ και οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία. Ο, ο εισηγητής μας, όπως ξέρουμε, είναι ο Μετίν Καζάκ. Και θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες και την ίδια την έκθεση. Να ξεκινήσουμε με την τροπολογία υπαριθμών 1. Πρώτη τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αρχή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να ελέγξουμε. Ε, δεν έχω την κάρτα, λέει κάποιος εκτός μικροφώνου, ούτε και εγώ λέει ο πρόεδρος θα ε, μετρήσω και τη δική μου ψήφο που είναι θετική. Το ελέγξαμε. Τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 3 και 4, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1. Υπάρχει αντίρρηση στην προφορική τροπολογία. Όχι. Να ψηφίσουμε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται. Διαδικαστικό εκτός μικροφώνου, δεν ακούμε. Δεν λειτουργεί η συσκευή μου και θα ήθελα να ψηφίσω υπέρ. Μπορείτε να μετακινηθείτε να χρησιμοποιήσετε άλλο, άλλη συσκευή. Να ξαναψηφίσουμε. Ψηφίζουμε την, ε, ελέγχουμε την ψηφοφορία της προφορικής τροπολογίας, υπάρχει μόνο ένα, αρχή της ψηφοφορίας, λήξη της ψηφοφορίας. Μπορέσατε να ψηφίσετε, κύριε Βάρτμουθ. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 7. Ε, έχει αποσυρθεί. Προφορική τροπολογία 2. Υπάρχει καμιά αντίρρηση στην προφορική αυτή τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Υπάρχουν 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπέρ 9. Υπέρ. Κατά χέρι απορρίπτεται 10 υπέρ κατά χέρι απορρίπτεται 12 υπέρ κατά χέρι απορρίπτεται 12 αρχή της ψηφοφορίας ελέγχουμε Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 17 καταπίπτει, 18 έχει αποσυρθεί. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 19 καταπίπτει. Η 15 καταπίπτει, λέει ο πρόεδρο. Προχωράμε στην ε, συμβαστική τροπολογία 3. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 27 υπέρ. 27. Οι άλλες ε, καταπίπτουν. 27 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 3 υπέρ. Όχι, συγγνώμη. Υπάρχει καμιά αντίρρηση στην προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται. 29 καταπίπτη, 31 καταπίπτει, 32 έχει αποσυρθεί, 30 καταπίπτει, 33 έχει αποσυρθεί, 34 έχει αποσυρθεί, 35. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε τροπολογία 36, αρχή της ψηφοφορίας. 36, αρχή της ψηφοφορίας. Και το αποτέλεσμα είναι ότι εγκρίνεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 38 υπέρ. 38 υπέρ. Η 37 ε, απορρίφθηκε. Να ελέγξουμε την 37 αρχή της πληροφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Το ίδιο ισχύει για τις 40 και 41. Εκτός μικροφώνου παρατήρηση δεν ακούσαμε. Ξέχασα να σας πω ότι ψηφίσαμε όχι μόνο τη 39 αλλά και την 40 και τη 41 ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα. Θέλετε να ελέγξουμε την ψηφοφορία. Εντάξει, ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά αρχή της ψηφοφορίας. 39, 40, 41. Τρεις τροπολογίες μαζί. Ελέγχουμε. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 43. 43. υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όλες οι άλλες καταπίπτουν μέχρι την συμβαστική τροπολογία 6. Ποιος είναι υπέρ, Κατά αποχές εγκρίνεται. Πενήντα έξι. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές εκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές εκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Απορρίφθηκε. 64. Να ελέγξουμε την ψηφοφορία για την 62, αρχή της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 64. Υπέρ, κατά, χέρι εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. χέρι εγκρίνεται. 67. Υπέρ. Κατά. χέρι απορρίπτεται. 68. Υπέρ. Κατά. χέρι εγκρίνεται. να ελέγξουμε την 68 αρχή της ψηφοφορίας. Ελέγχουμε την ψηφοφορία για την 68 αρχή της ψηφοφορίας. The And it was adopted. Εγκρίνεται. Amendment number 9. Ε, συμβαστική τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται, συγγνώμη. Ε, συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Ε, αποχές εγκρίνεται. Προχωράμε στην 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική τροπολογία 11. Υπέρ. Να προσθέσουμε μια λέξη relevant member states, ε, τα, σχετικά κράτη-μέλη στην συμβαστική τροπολογία 11. Υπάρχει καμιά αντίρρηση στην ε, προφορική τροπολογία. Μία λέξη μόνο προσθέτουμε. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Να ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία με την, ε, τη συμβαστική τροπολογία με την προφορική αυτή τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Γιάννη But, but you, you object the amendment? Okay. Then we vote as it is. Υπάρχει αντίρρηση στην προφορική τροπολογία, τότε να ψηφίσουμε τη συμβαστική τροπολογία ως έχει, χωρίς την προφορική τροποποίηση. Συμβαστική τροπολογία 11, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 12. Την 84. Ναι, διότι 83 απορρίφθηκε. 84. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 84 ψηφίζουμε. Θα ξαναψηφίσουμε. Καταπίπτει λοιπόν η τροπολογία 84. Α, εντάξει, σύμφωνοι. Ναι, διότι απορρίφθηκε η 83, γι' αυτό πρέπει να ψηφίσουμε την 84 και αυτό ξανακάνουμε. Ψηφίζουμε την 84, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 85. Είναι συμβατή με τη συμβαστική τροπολογία 12. Ψηφίζουμε τροπολογία 85 υπέρ. Τροπολογία 85. Όχι, δεν καταπίπτει. Υπέρ της τροπολογίας 85. Ήδη ψηφίσαμε τη συμβαστική τροπολογία, την 12. Την εγκρίναμε. Ψηφίζουμε την τροπολογία 85. Μία λέξη αλλάζει. Άρα πρόκειται για τροπολογία. Υπέρ, κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Αρχή της ψηφοφορίας. 85. Αρχή της ψηφοφορίας. Uh, the vote Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Προχωράμε στην 92. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τη τελική ψηφοφορία Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Open. The vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. και στους κοιόδεις εισηγητές φυσικά. Ας προχωρήσουμε τώρα.

ψηφίσουμε την έκθεση υπαριθμών 10, το σημείο 10, μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Έγκριση τροπολογιών. Η συγητής Γιούλιου Βίνκλερ. Έχουμε πέντε τροπολογίες. Και σήμερα θα ψηφίσουμε μόνο τις τροπολογίες. Την έκθεση θα την ψηφίσουμε τον Αύγουστο. Να προχωρήσουμε λοιπόν. Πέντε τροπολογίες του εισηγητή. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί, on block? Υπάρχει καμιά αντίρρηση στο να ψηφίσουμε μαζί και τις πέντε τροπολογίες.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 και ακολουθούμε την ε, πρόταση του εισηγητή να ξεκινήσει ένας άτυπος τριμερής διάλογος με στόχο την επίτευξη συμφωνίας ε, στην πρώτη ανάγνωση. Γι' αυτό προτείνω να ε, λάβουμε την εξή απόφαση σύμφωνα με του ε, διαδικαστικού ε, κανόνε τη ε, Επιτροπή ΣΥΝΤΕ. Να ξεκινήσουμε άτυπε διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο και την Κομισιόν, να πετύχουμε συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση και κατόπιν οι τροπολογίε που υιοθετήσαμε θα, αποτελέσουν, τη βάση για την εντολή τη διαπραγματεύτική ομάδα, η οποία θα αποτελείται από τον εισηγητή μα, Γιούγλιου Βίνκλερ, και του κοιόδη εισηγητέ, Κούτα, Σόλτ και Ζαραντή. Συμφωνείτε με την πρόταση αυτή, υπάρχει καμία αντίρρηση. Εγκρίνεται λοιπόν. Να προχωρήσουμε τώρα στο σημείο 3 στην ημερήσια διάταξη, το οποίο δεν κάναμε χθες, διότι η συνάδελφός μας, η κυρία Μουσκαρδίνη, δεν ήταν εδώ σήμερα στην αρχή της συνεδρίασης. Όπως θα γνωρίζετε, το θέμα αυτό έχει να κάνει με την ένδειξη της χώρας καταγωγής. Καταγωγή λοιπόν. Δεν έχουμε διακοπές ακόμα, παρακαλώ. Την επόμενη Παρασκευή, σας παρακαλώ. Την επόμενη Παρασκευή ξεκινάνε διακοπές, την προσοχή σας παρακαλώ. Και θα παρακαλούσα τους μη βουλευτές να μην συζητάνε τόσες αιθούσεις. This applies to everyone. This is not a forum, a public forum. So, let's go back to our... Ας ε, επανέλθουμε λοιπόν στην ε, δουλειά μας. Το σημείο 3 είναι εξέταση σχεδίου έκθεσης της Κριστιάνας Μουσκαρδίνη για την ένδειξη της χώρας προέλευσης σε ορισμένα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες. Όπως θα γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κάποιο κανονισμό που να ισχύει σε εξαγωγής από τρίτες χώρες ε, σχετικά με την ε, ένδειξη της χώρας καταγωγή στα προϊόντα και αυτό πιθανότατα να έχει να κάνει με την έλλειψη αυτό μπορεί να οδηγεί σε ε, έλλειψη πληροφόρησης των Ευρωπαίων καταναλωτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υιοθετήσει με μεγάλη πλειοψηφία ε, σχετική πρόταση. Σήμερα εξετάζουμε το σχέδιο έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού. Δίνω λοιπόν το λόγο στη συναδελφό μας την Κριστιάνα Μουσκαρδίνη. Παρακαλώ. Grazie <coughs> Presidente, come i colleghi sanno abbiamo già avuto modo due volte di, avere in Εμείς για δύο φορές ανταλλάξαμε απόψεις για το θέμα και όπως ε, θύμισε και ο Πρόεδρος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ολομέλεια ε, κατάφεραν να εκφραστούν και να πούνε ότι χρειάζεται ένας κανονισμός ούτως ώστε να τεθεί στο ίδιο επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις άλλες χώρες ανταγωνιστές. Βέβαια αυτή η πρόταση χρειάστηκε ορισμένες τροπολογίες. Διότι ναι μεν όλος ο κορμός παραμένει επίκαιρος, ε, υπό το φως των διαφόρων γεγονότων της τελευταίας πενταετίας, χρειάζεται ορισμένες βελτιώσεις και τροπολογίες για να εξηγήσουμε καλύτερα τα πράγματα και για να μπούμε στην ουσία των πραγμάτων. Σήμερα, ακριβώς επειδή έχουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας η οποία δίνει συναποφασιστική αρμοδιότητα στο Κοινοβούλιο και μεγαλύτερες πολιτικές εξουσίες, χρειάστηκε να παρουσιάσουμε μία τροπολογία που να λέει οποιαδήποτε τροπολογία του κανονισμού που θα εγκριθεί κάποια στιγμή, δηλαδή οποιαδήποτε προσθήκη κατηγοριών ή κατάργηση ε, κατηγοριών θα πρέπει να περάσει από το Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε να την εγκρίνουμε, να εγκρίνουμε δηλαδή αυτή την πρόταση τροπολογίας κομισιών. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την Κομισιόν. Ε, εμείς θα πρέπει σήμερα να αξιολογήσουμε το γενικό κορμό, δηλαδή τη σκαλωσιά του κανονισμού και να κάνουμε μια γενικότερη εξέταση των τροπολογιών, να ακούσουμε και άλλες τροπολογίες που εσείς θα θεωρήσετε σωστές και να το συζητήσουμε το θέμα ολοκληρωτικά τον Σεπτέμβριο. 30 Αυγούστου λίγη κατάθεση τροπολογιών. Ελπίζω λοιπόν ότι θα καταφέρουμε από κοινού να συνεχίσουμε τη δουλειά μας η οποία ήταν ιδιαίτερα επωφελής για την ανταλλαγή απόψεων και λόγω φυσικά της βοήθειας του καθενός από εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είχαμε ένα πρώτο έγγραφο εργασίας από την κυρία Μουσκαρντίνη. Πλέον ε, έχουμε το ε, σχέδιο έκθεσης. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ο Τζανλούκα Σούστα, πολύ σύντομα. Την πολιτική μας αντιπαράθεση για το θέμα την, είχαμε στο, ε, την έχουμε ήδη κάνει Εμείς θα πρέπει να διαφυλάξουμε δύο αρχές. Πρώτον, το ελεύθερο εμπόριο ως μέσο για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Πρέπει όμως να επαναλάβουμε το θέμα της αρχής της προστασίας των ελευθέρων ανταλλαγών είναι φυσικά αν οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Κίνα, η Ινδία έχουν ένα νομικό μέσο αντίστοιχο με αυτό και εμείς δεν το έχουμε, ε, τότε φυσικά και εμείς το χρειαζόμαστε. Και αυτό θέλει δηλαδή και ο κανονισμός, αυτό θέλει και η έκθεση της ε, κυρίας Μουσκαρδίνη, την οποία ευχαριστώ. Και οι τροπολογίες που κατατέθηκαν πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση διότι θέλουν την προστασία του καταναλωτή που είναι και η σωστή προσέγγιση του προβλήματος Θέλουν επίσης να καλύψουν και άλλες ελλείψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλους τομείς. Είπαμε προστασία λοιπόν των καταναλωτών και μετά καταπολέμηση της απομίμησης. Διότι Σκεφτείτε τι γίνεται με τις απομιμήσεις, απομιμήσεις ε, εντάξει σε προϊόντα ανόητα όπως είναι δεν ξέρω τι τα φρουφρού και τα παπούτσια αλλά πόσο είναι επικίνδυνες αυτές οι απομιμήσεις όταν φύγουν τον τομέα των φαρμάκων που είναι πολύ πιο ουσιαστικός. Λοιπόν, και αυτή η πλευρά είναι πολύ σημαντική και ξέρουμε ότι εδώ πρόκειται για κανονισμό, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δεσμευτικός για τα κράτη-μέλη. Χρειάζεται ίσως ε, κάποια λεξική διόρθωση το κείμενο, αλλά πάει προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ζαντό. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Υποστηρίζω την έκθεση της κυρίας Μουσκαρδίνη. Είναι πολύ σημαντική. Η προσέγγιση είναι πολύ πιο περιοριστική από αυτή του Συμβουλίου. Δύο πράγματα όμως στην έκθεση ανακατεύεται ε, το made in μαζί με το κοινωνικό και το περιβαλλοντικό πακέτο. Δεν ξέρω, θα έπρεπε να μην μπερδεύουμε το πού έχει κατασκευαστεί το προϊόν με την μέθοδο παραγωγής του προϊόντος. Θεωρούμε λοιπόν ότι το κοινωνικό και περιβαλλοντικό λάμπελ είναι διαφορετικό πράγμα και δεν πρέπει να το μπερδεύουμε με την προέλευση. <coughs> Ίσως θα, θέσουμε και μία πρωτοβουλία, ε, τροπολογία συγγνώμη, για το πώς προβάλλει η εισηγήτρια τα ευρωπαϊκά προϊόντα και πώς προβάλλει τα εισαγόμενα προϊόντα. Δηλαδή εμάς δεν μας αρέσει αυτό. Τι η άποψη το ότι τα δικά μας προϊόντα είναι καλά και αυτά που έρχονται απ' έξω δεν είναι. Σίγουρα να γράφεται η προέλευση του προϊόντος, αλλά καμία κρίση για αυτή την προέλευση. Οι σκιώδεις εισηγητές θέλουν να πάρουν το λόγο από τους φιλελεύθερους. Ο Νικόλο Ρινάλντι. Υποστηρίζουμε αυτήν την έκθεση και την θέση της Κριστιάνα Μουσκαρδίνη. Οι προλαλήσαντες τα πανόλα αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό αυτή η έκθεση και στο μέλλον δηλαδή ε, έναντι του Συμβουλίου να αποτελεί λέση τμήμα μίας πιο ολοκληρωμένης ε, ε, στρατηγικής. Διότι εδώ εμείς πρέπει να επιβεβαιώσουμε την αρχή ότι όχι μόνο εμείς ε, θέλουμε να βοηθήσουμε την οικονομία μας προστατεύοντας το δικό μας know-how το παραδοσιακό know-how, αλλά επίσης γιατί τονίζουμε και αυτήν την αρχή της αμοιβαιότητας η οποία χρειάζεται στην αγορά και άλλοι είναι πρικολικισμένοι με τέτοιου είδους κανόνες η Κίνα, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ινδία και εμείς λόγω δικής μας επιλογής ακόμη δεν το είχαμε. Συμφωνώ με τον Ζαντό όταν λέει ότι θα πρέπει να αποφύγουμε η σήμανση να γίνει η, να γίνει η ετικετοποίηση του καλού μαθητή, του πρώτου μαθητή της τάξης, δηλαδή αυτού, ότι τα δικά μας προϊόντα είναι τα καλύτερα προϊόντα και των αλλωνών δεν είναι. Τα προϊόντα μας λοιπόν θα, θα πρέπει να έχουν τη σήμανση κατασκευασμένα στην Ευρώπη. Και μετά για την τροπολογία 6. Πρόκειται για μια ανησυχία που μας εξέφρασε σαν οι επιχειρηματίες σχετικά με την ε, γραφειοκρατική επιβάρυνση που, θα μπορεί, να επιφέρει η σήμανση. Και αυτό το λέει φυσικά και η συγκήτρια ότι η σήμανση δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί με επιπλέον γραφειοκρατική φόρτιση αλλά θα πρέπει νομίζω να συμπληρωθεί, να πούμε κάτι παραπάνω γι' αυτό. Δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Μία που επηρεάζει το εμπόριο και τις εμπορικές συναλλαγές και μια άλλη η οποία είναι πολύ περισσότερο επί της ουσίας, ουσιαστικά έχει να κάνει και με τις α, πολιτικές ελευθερίες. Λέγεται στο κείμενο ότι θέλουμε να δούμε ποια είναι η δικαιοδοσία αυτή η οποία μπορεί να αποφασίσει σε περίπτωση διαφοράς, δικαστικής διαφοράς. οι, τα περισσότερα, οι περισσότερες εμπορικές συμβάσεις λένε σε περίπτωση διαφοράς η διαφορά αυτή θα πρέπει να διευθετηθεί σύμφωνα με το Βρετανικό δίκαιο. Και αυτό είναι ιδιαίτερα η αναφορά αυτή στο Βρετανικό δίκαιο όσον αφορά τις συμβάσεις διεθνούς εμπορίου είναι ιδιαίτερα επωφελής στις, στα συμβαλώμενα μέρη. Διαφορετικά δεν επρόκειτο ποτέ να συμφωνήσουμε για ποια σύμβαση. Ανησυχώ λοιπόν πολύ που βλέπω εδώ πέρα την αναφορά που γίνεται στην αρμόδια δικαιοδοσία. Ουσιαστικά αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε εδώ πέρα είναι ότι τα συμβαλώμενα μέρη θα μπορούν να επιλέγουν τη δικαιοδοσία στην οποία θα υπαχθούν και μάλλον το δικαίωμα αυτό να επιλέξουν δεν θα υπάρχει πλέον, θα τους αποσυρθεί. Θα ήθελα εγώ να αντιταχθώ σε κάτι τέτοιο και ελπίζω ότι και οι υπόλοιπες πολιτικές ομάδες θα συμφωνήσουν μαζί μου. Να δούμε δηλαδή ξεκάθαρα πώς έχει η κατάσταση και να δώσουμε στα συμβαλόμενα μέρη τη δυνατότητα να επιλέξουν τη δικαιοδοσία στην οποία θέλουν να υπαχθούν. Ενδεχομένως τώρα να βγω από το πεδίο αρμοδιότητας της δικής μας επιτροπής, γιατί δεν θα μιλήσω άμεσα για το θέμα του εμπορίου. Είμαστε όλοι βουλευτές και πολίτες των χωρών μας και θα ήθελα να αφαιρθώ σε ένα άλλο σημείο. Διαδικασία εναρμόνισης της νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα επωφελές. Λέγεται επίσης στο σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος Στοχόλμη στην εισαγωγή ότι οι άνδρες και οι γυναίκες στην Ευρώπη θέλουν να ζουν σε μια ευήμερη ειρηνική Ευρωπαϊκή Ένωση όπου θα παρέχονται όλες οι συνθήκες ασφάλειας. Αυτό αληθεύει. Αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι στην προσπάθεια εναρμόνισης που γίνεται, η οποία δεν διεξάγεται σωστά, έχουμε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης οι συνέπειες αυτού είναι ιδιαίτερα επιζήμιες για τα συμφέροντα των Βρετανών πολιτών και δύο πολίτες από τη δική μου εκλογική περιφέρεια κατέληξαν στη φυλακή στην Ουγγαρία. Λυπάμαι που ο κύριο Στάνση δεν είναι στην αίθουσα. Εκατό μέρες πέρασαν στη φυλακή στην Ουγγαρία περιμένοντας να δικαστούν και θα μπορούσαν να είχαν μέχρι και τρία χρόνια στη φυλακή περιμένοντας να γίνει δίκη. Οι Ουγγρικές αρχές τους φέρθηκαν πολύ σωστά και τελικά τους απελευθέρωσαν, μολονότι οι κατηγορίες εναντίον τους εξακολουθούν να υφίστανται. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι δεν είναι ίδια όλα τα νομικά συστήματα τα οποία ισχύουν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένα νομικά συστήματα σε, σε ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ένα υψηλό επίπεδο προστασία, το habeas corpus για παράδειγμα, και μια τέτοια χώρα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Το να προσπαθούμε όμω να εναρμονίσουμε όλα αυτά τα νομικά και δικαστικά συστήματα θα οδηγήσει σε μείωση των δικαιωμάτων των πολιτών, θα μειώσει την ασφαλειά τους, θα μειώσει το επίπεδο δικαιοσύνης, ουσιαστικά θα θέσει εν κινδύνο την ίδια την ελευθερία τους. Επομένως θα θέλω να ζητήσω από τους βουλευτές, από τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες και κυρίως από την αριστερά, αλλά και απευθύνομαι στους ε, βουλευτές των φιλελευθέρων, να έχουν κατά νου το εξή η εναρμόνιση όταν δεν είναι καλά σχεδιασμένη, όπως συμβαίνει ακριβώς το πρόγραμμα της Στοκόλμης, ουσιαστικά αντιτίθεται στα δικαιώματα του πολίτη. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, με συγχωρείτε. Ο κύριο Σόλτ πρώτα έχει το λόγο. Σα ξέχασα και στη συνέχεια προφανώ θα πάρει το λόγο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Ήθελα να σας δώσω τη βασική μας θέση. Συμμεριζόμαστε τη βασική θέση της έκθεσης αυτής. Ευχαριστούμε και τη δουλειά που έχει γίνει όσον αφορά αυτό που μόλις υπόθηκε και από τον συνάδελφο Ρινάλντι. είναι ότι ε, ο επιχειρηματικός κόσμος στις τελευταίες εβδομάδες ε, κοιτάει με τρόμο τα γραφειοκρατικά βήματα που γίνονται για να γίνει το σύστημα αυτό διαφανές. Ε, φοβούνται ότι μπορεί να αυξηθούν ραγδαία οι δαπάνες παραγωγής το κόστος παραγωγής. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε το εκτιμώντας ε, μήπως μπορούμε να το ε, διατυπώσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια για να διασκεδάσουμε τις ανησυχίες που υπάρχουν. ε, ίσως να υποβάλουμε σχετική τροπολογία. Κατά τα άλλα, ευχαριστούμε τη δουλειά που έχει γίνει. I call on commission to take the floor. Η Κομισιόν να πάρει το λόγο, παρακαλώ. Thank you, Chairman. And thank you to the rapporteur uh, and... Uh, Ευχαριστώ τον εισηγητή και την Επιτροπή για τη δουλειά που έγινε. Γενικά συνεμεριζόμαστε όπως γνωρίζετε. Ε, τη θέση του εισηγητή για τις ε, τροπολογίες που έχει υποβάλει. Το έχουμε συζητήσει αυτό νωρίτερα. Ε, ε, τώρα με τη συνθήκη της Λισαβόνες μπορούμε να εφαρμόσουμε τις πράξεις κατεξουδότηση για να έχουμε καλύτερη ισορροπία όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Κομισιόν θέλουμε λοιπόν, ε, όσον αφορά τι αρμοδίε ε, της Κομισιόν, να τροποποιεί το ε, παράρτημα. Θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή κατά την εφαρμογή των τεχνικών κανονισμών. Οι εισαγωγή μας και η έμποροι μας δεν ε, φέρουν ε, σημαντικό ε, διοικητικό άχθος όσον αφορά την επισήμανση της προέλευσης και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα. Συμμεριζόμαστε τη θέση ότι η προέλευση είναι ξεχωριστή πληροφορία και πρέπει να λαμβάνει απλά ο καταναλωτής πληροφορία σχετικά με την προέλευση του προϊόντος. Υπάρχει μια τροπολογία την οποία δεν έχουμε συζητήσει νωρίτερα και για την οποία η Κομισιόν θα πρέπει να προχωρήσει περισσότερο εις βάθος. Δεν είχαμε το χρόνο ακόμα να υποβάλουμε στην νομική μας υπηρεσία το σύνολο των τροπολογιών ώστε να έχετε πιο αναλυτική θέση της Κομισιόν. Υπάρχει τροπολογία στην οποία ο συγητής λέει ότι η Κομισιόν θα πρέπει να εξασφαλίσει ένα ελάχιστο επίπεδο εναρμόνισης όσον αφορά το σύστημα κυρώσεων στα κράτη-μέλη. θα πρέπει να δούμε τι χρειάζεται, τι είδους ε, ρύθμιση χρειάζεται από πλευράς της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ και πάλι. Μήπως θα μπορούσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν να ε, απαντήσει στις ε, δύο ερωτήσεις που έκανα. Εάν δεν μπορεί να το κάνει αυτό, μήπως μπορώ να στείλω επιστολή, να λάβω ε, γραπτή απάντηση. Δεν προσπαθήσατε καν, αγνώρισατε τελείως ερωτήσεις μας και είναι πολύ σημαντικά τα δύο αυτά σημεία. Θα απαντήσει η Κομισιόν στις συγκεκριμένες ερωτήσεις που τέθηκαν. honest, uh, uh, the... Για να είμαι ειλικρινής δεν κατάλαβα τι σχέση έχει η ερώτησή σα με τον κανονισμό που έχουμε. Ήταν πολύ πολιτική ερώτηση, είχε να κάνει με την εναρμόνιση. Ρώτησα επίσης σχετικά με το, τα δικαιώματα των συμβαλωμένων ε, σε εμπορικές συμφωνίες να επιλέξουν ε, την ε, δικαιοδοσία που θα ορίζει τις τις συμφωνίε του. 90 ε, δευτερόλεπτα μίλησα, 1,5 λεπτό μίλησα για το θέμα αυτό. Ναι, αλλά δεν υπάρχει τίποτα στον κανονισμό αυτό που έχει να κάνει με διεθνείς συμβάσεις ε, ή διαφωνίε. Ανέφερα το σημείο εκεί που, λέμε το, ε, εκεί που μιλάμε για τη δικαιοδοσία που είναι υπεύθυνη για την επίλυση κάποια συγκεκριμένη διαμάχη. Για αυτό το πράγμα ήθελα να διευκρινίσω Καλά, πτώση διαδικαστικό όμω. Νομίζω ότι υπάρχει μια παρανόηση εδώ πέρα. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος θα αναφέρεται εδώ πέρα σε ένα άλλο κείμενο, στο οποίο θα μπορούσαμε όντω να κάνουμε τι παρατηρήσει αυτέ. η παρατηρήση έχει να κάνει με το πρόγραμμα τη Στοκχόλμη όμω, και δεν σχετίζεται με τον κανονισμό για την ένδειξη χώρα προέλευση για το οποίο μιλάμε. Το δικό σου επιχείρημα είναι σίγουρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό το λόγο θα πρότεινα να αποστείλετε μία γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το συγκεκριμένο όμως ζήτημα του προγράμματος της Στοκχόλμης. Γιατί το ερώτημά σας με το πρόγραμμα αυτό σχετίζεται και όχι με τον κανονισμό που συζητάμε σήμερα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ειλικρινά όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην εργασία που κάναμε, τους σκιώδεις συγητές αλλά και τους υπόλοιπους συναδέλφους που τους τελευταίους μήνες είχαν ε, την ευγένεια να κάνουν προτάσεις και να συζητήσουν μαζί μου για τις διάφορες πτυχές του ζητήματος. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μία ακόμη φορά κατέδειξε ότι πέρα από τους διαχωρισμούς που μπορούν να υπάρχουν ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες, έχει και μια κοινή πολιτική βούληση προκειμένου να βοηθήσει τους Ευρωπαίους πολίτες και να καταλήξει σε κανονισμούς οι οποίοι ακολουθούν ένα κοινό μέτωπο, έχουν μια κοινή γραμμή. Όλοι αυτοί οι κανονισμοί, το ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σαφής και εμφανής ετικετοθεσία, όλα τα ζητήματα αυτά που έχουν να κάνουν με την ένδειξη της χώρας προέλευσης. Όλες οι περιβαλλοντικές πτυχές του ζητήματος που θίξατε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, νομίζω ότι είναι στοιχεία τα οποία θα αντικατοπτρίζονται και στις τροπολογίες που θα υποβάλουν οι συνάδελφοι, τροπολογίες με τις οποίες θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο το κείμενο. Επίσης είναι πολύ σημαντικό το ότι καταφέραμε να καταλήξουμε σε μία τοποθέτηση που μας επιτρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να πούμε στο Συμβούλιο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις νέες του αρμοδιότητες προσπαθεί να βρει λογικούς συμβιβασμούς αλλά παράλληλα δεν έχει την πρόθεση να κάνει πολύ μεγάλες εκχωρήσεις ή να υποχωρήσει σε ζητήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και ζητήματα για τα οποία πολλές φορές το Συμβούλιο αφήνει να περάει χρόνος χωρίς να προσπαθεί να βρει άμεσα λύση. Ευχαριστώ. Yes, and, uh, Ο κύριος Φιέλνερ ζήτησε το λόγο. Καταρχήν θα ήθελα ε, να πω όσον αφορά τη συζήτηση αυτή. Δυστυχώς έπρεπε να πάω στην ε, ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, για να ψηφίσω εκεί. Θα ήθελα όμως να προσθέσω κάτι. Όπως ξέρετε αρκετοί από εσά εδώ πέρα, εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα αυτό. Είμαι αρκετά σκεπτικός απέναντι στην πρόταση. Ε, μόνος μου έχω υποβάλει πρόταση που να διασφαλίζει το να μην γράφουν αναλήθειες οι παραγωγοί. Ε, και για να καταπολεμήσουμε ε, ε, αθέμητες μεθόδους διάθεση στην αγορά. Έχουμε διαφορετικά σημεία κίνηση εγώ και ο εισηγητής, ωστόσο πιστεύω ότι είναι πολύ ισορροπημένη η πρόταση που υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες είναι πολύ καλή. Στις δικές μου τροπολογίες θα επικεντρωθώ στο πεδίο εφαρμογής, ποια προϊόντα θα καλύπτονται και ποια όχι. Και θα εξετάσουμε επίσης ποιο, τι, είδου ε, ορισμό ε, για την ε, χώρα προέλευσης θα χρησιμοποιήσουμε. Αλλά όπως σας είπα, είναι διαφορετικά τα σημεία κίνησής μας, αλλά είχαμε πολύ καλή συνεργασία και ελπίζω ότι θα συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Ευχαριστώ. It was also clarified that Ε, επίσης ξεκαθαρίσαμε ότι αυτό που είπε ο William Dartmouth δεν έχει καμία σχέση με το θέμα αυτό. Ε, είχε να κάνει με το σημείο 11 το οποίο συζητήσαμε χθε. Να σας ενημερώσω ότι η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες είναι 30 Αυγούστου. Since uh, uh, Καθότι η συνάδελφός μας Κουίσχαουτ Ρόβολ δεν είναι παρούσα, καταφθάνει όμως, ας προχωρήσουμε. Με ενημερώνω ότι θα φτάσει σε δύο λεπτά.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 Willem Dartmouth. He's there. Could you move to Uh, William Dartmouth, are you ready? Ε, William Dartmouth, είσαστε έτοιμος να ε, μας μιλήσετε για το σημείο 13. Καθότι έφτασε ο William Dartmouth, θα προχωρήσουμε στο σημείο 13, εν αναμονή της κυρίας Κουίστχαουτ Ρόβολτ, να φτάσει στην αίθουσά μας. Σημείο 13 λοιπόν. Πρόκειται για πρώτη ανταλλαγή απόψεων. για το θέμα της χορήγησης εγγύησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγύησης για σχέδια εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας παρακαλώ, μην έχετε συζητήσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών μας. Since, um, Has arrived. Έφτασε η κυρία Κουίστχαρτ Ρόβολ. Ας προχωρήσουμε λοιπόν. Ας πάμε πίσω, δηλαδή στο σημείο 12. Ευρωπαϊκή Ένωση, Γεωργία και Διεθνές Εμπόριο. Όπω ξέρετε, η Επιτροπή Άγκρη ετοιμάζει έκθεση πρωτοβουλία για τη Γεωργία και το Διεθνές Εμπόριο, η οποία θα ε, καλύπτει μια σειρά από θέματα που έχουν να κάνουν με το εμπόριο, που εμπίπτουν στι αρμοδιότητες της Επιτροπής μας. Γι' αυτό η ΙΝΤΕ συντάσσει γνωμοδότηση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 σε απόλυτους αριθμούς δεν φαίνεται να ε, καλύπτει ε, τόσο μεγάλο μερίδιο των ε, εμπορικών συναλλαγών. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, αλλά συμφωνούμε ότι το εμπόριο των γεωργικών προϊόντων είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό θα πρέπει η Επιτροπή μας να είναι μια συνδεδεμένη Επιτροπή στην έκθεση αυτή και όχι απλά να γνωμοδοτήσει. Υπάρχει συμφωνία όμως σχετικά με αυτό με τον εισηγητή. Υπάρχει συμφωνία σχετικά με το ποιο θα κάνει τι και θα ήθελα καταρχήν εδώ με τους συναδέλφους ε, εντό της Επιτροπής μας αλλά φυσικά και με τους συναδέλφους της Επιτροπής Γεωργίας να έχω συζητήσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών. Η κατάσταση είναι εξή από πλευράς της Ευρώπης. Ε, μπροστά μας έχουμε το μέλλον της ε, ε, κοινή γεωργικής πολιτικής και στα πλαίσια του ΠΟΕ περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον του γύρου της Δόχα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι θέλουμε από πολιτικής πλευράς, αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερον, Ε, κάνουμε ένα σωρό, συνάπτουμε ένα σωρό ε, εμπορικές συμφωνίες, ε, GPS, FTS κλπ, οι οποίες έχουν επιπτώσεις στις γεωργικές αγορές, στους υπεύθυνους χώρους της Ευρώπης, θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό και γι' αυτό θα πρέπει να αποτελούν κομμάτι της έκθεσης αυτής. Επίσης ε, κάτι που θα συζητήσουμε περαιτέρω είναι αυτό. Πρώτο σχέδιο της έκθεσης ε, θα υποβληθεί το φθινόπωρο, μάλλον τον Οκτώβριο και στόχος της Επιτροπής Γεωργίας είναι να πάμε στην Ολομέλεια αρχές του 2011. Ε, μπορεί να σας φαίνεται μεγάλο το χρονικό διάστημα αυτό, καθότι όμως θα πρέπει να επικεντρωθεί η δουλειά μας ε, στους πρώτους που θα, συ, που θα σημειωθούν ε, όσον αφορά το ε, μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής. νομίζω ότι είναι πολύ ρεαλιστικό το χρονοδιάγραμμα. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την σίγουρα καλή συνεργασία που θα έχουμε και σας ευχαριστώ για την ε, προσοχή σας και πάνω απ' όλα καλές διακοπές. Εγώ σχεδόν έχω φύγει ήδη. Μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση. Υπάρχει κάποιος που θα θέλει το λόγο. Για το ζήτημα αυτό υπάρχουν παρατηρήσεις, παρεμβάσεις σε σχέση με την γνωμοδότηση που θα συντάξει στην αδελφός μας. Παρακαλώ. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Νόμιζα ότι οι μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες θα έπαιρναν το λόγο πρώτες. Θα ήθελα να κάνω μια-δυο γενικές παρατηρήσεις καταρχάς. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε Οποιαδήποτε, οποιαδήποτε έκθεση υποβάλλεται όσον αφορά το διεθνές εμπόριο και τη γεωργία, προκειμένου να εξετάσουμε καλύτερα τις βασικές αρχές που διέπουν την οργάνωση της γεωργίας. Στην Ευρώπη, καταρχάς και στη συνέχεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Προφανώ η γεωργία, τα γεωργικά προϊόντα αποτελούν πολύ μεγάλο τμήμα των εμπορικών συναλλαγών. Κατά την άποψή μου πιστεύω ότι θα πρέπει να επιστρέψουμε στι αρχικέ βασικέ αρχέ. Η γεωργία πρέπει να έχει κυρίω ω στόχο να παράγει τρόφιμα προκειμένου να μπορούν να τρέφονται οι άνθρωποι και μια γεωργική πολιτική σε ένα πολιτισμένο κόσμο θα πρέπει να έχει ως στόχο την διατροφή των ανθρώπων. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποσυτίζονται ακόμα και θα πρέπει αυτό να γίνεται με έναν τρόπο που να σέβεται και να προστατεύει το περιβάλλον. Δυστυχώς στον καπιταλιστικό κόσμο που υφίσταται, που υπάρχει, η προτεραιότητα της α, διατροφής των ανθρώπων δεν υφίσταται. Προτεραιότητα είναι οι τιμές, οι γεωργικές τιμές και το κέρδος και αυτό ουσιαστικά διέπει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται το εμπόριο στα γεωργικά προϊόντα. Και βλέπετε τα αποτελέσματα σε παγκόσμιο επίπεδο της τακτικής αυτής. Ζούμε ακόμα μια απίστευτη κατάσταση όπου υπάρχουν εκατοντάδες, εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι υποσυτίζονται, υπάρχουν παιδιά τα οποία πεθαίνουν από τη φτώχεια και την ένδυα. Πήγα σε μια περιοχή της Βραζιλίας πριν από μερικά χρόνια. Όταν ήμουν εκεί έμαθα για ένα τεράστιο σκάνδαλο. Υπήρχαν ε, παιδιά αυτοχθόνων τα οποία πέθαιναν από υποσιτισμό στα χωριά τους και δίπλα στα χωριά αυτά βλέπατε κτήματα, εκτροφία με τα πιο ε, παχιά ζώα που θα μπορούσε ποτέ να δει κανείς. Η κατάσταση αυτή όμως δεν επικεντρώνεται μόνο στη χώρα αυτή, αλλά είναι γενικευμένη. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να αναδιοργανωθεί ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται και διεξάγεται το εμπόριο σε γεωργικά προϊόντα. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιφάσεις στον τρόπο με τον οποίο τα πράγματα οργανώνονται αυτή τη στιγμή. Στο Δουβλίνο, για παράδειγμα, βλέπουμε προϊόντα τα οποία έρχονται από το Ισραήλ ή από την Κύπρο, Βλέπουμε ότι ε, υπάρχουν πάρα πολλά αεροπλάνα, γίνονται πάρα πολλές πτήσεις οι οποίες μεταφέρουν ε, τρόφιμα από τη μία χώρα στην άλλη, ενώ αν τα πράγματα είχαν, ε, οργανωθεί διαφορετικά με πολύ πιο λογικό τρόπο, θα μπορούσαμε να είχαμε πιο τοπική παραγωγή, η οποία θα ήταν και πιο φιλική για το περιβάλλον. Έχουμε επίση και το ζήτημα των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων, κυρίως όσον αφορά τους ε, σπόρους ε, και όσον αφορά κάποιες βασικές ε, καλλιέργειες. Νομίζω ότι τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα μπορούν να είναι ιδιαίτερα επιζήμια για το περιβάλλον και να έχουν πάρα πολλούς, πάρα κινδύνους. Υπάρχουν μεγάλες εταιρείες, πολλές φορές εταιρείες παραγωγής χημικών προϊόντων που προκειμένου να δώσουν περισσότερα χρήματα και μεγαλύτερα μερίσματα στους μετόχους τους προχωρούν σε γενετική τροποποίηση σε πάρα πολλούς σπόρους, αλλά και σε βασικά τρόφιμα όπως το ρύζι. Και γνωρίζουμε μετά από πειράματα τα οποία έχουν γίνει ότι η γενετικά τροποποιημένοι σπόροι θα συμπεριφερθούν υποτίθεται με έναν τρόπο πολύ προβλεπόμενο. Στην πράξη όμως δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν οι σπόροι αυτοί, πώς θα επηρεαστούν από τις κλιματικές αλλαγές. Και αν θέλετε όλο το κεφάλαιο σπόρων ολόκληρων χωρών και περιοχών θα μπορούσε να τεθεί εν κινδύνο. Και αυτό πάλι βέβαια γίνεται προκειμένου να αποφεληθούν οι μεγάλες εταιρείες και όχι για να αποφεληθούν οι πληθυσμοί της Ευρώπης, της Ινδίας ή άλλων περιοχών του κόσμου. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι θα πρέπει να εστιαστούμε στα σημεία αυτά, θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας να δούμε ποια είναι τα θεμελιώδη κριτήρια τα οποία θα πρέπει να ισχύουν. Συγκεκριμένα ότι η γεωργία θα πρέπει να υφίσταται για την ευημερία του ανθρωπίνου είδους και όχι για να γίνονται πιο πλούσιοι οι μέτοχοι κάποιων μεγάλων εταιριών. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, υπάρχουν άλλοι που θα θέλουν το λόγο. Κύριος Ράντολφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συνεχίσω τον ίδιο συλλογισμό του συναδέλφου Higgins. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι η επιστημιστική κατάσταση στον κόσμο χειροτερεύει. Χειροτερεύει εδώ και πολλά χρόνια. Μέχρι το 2002-2003 η κατάσταση στις τρίτες χώρες ήταν καλύτερη σε σχέση με τη δεκαετία του 60, ενώ τώρα ο συνολικός αριθμός ανθρώπων ε, που ε, υποσυτίζονται μεγαλώνει. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Αντιμετωπίζουμε και την παγκοσμιοποίηση των ε, καταναλωτικών συνηθιών σε όλο τον κόσμο. Το βλέπουμε αυτό και με την κατανάλωση κρέατος. Η μετάβαση προς την μεγαλύτερη κατανάλωση κρέατος ε, έχει αυξηθεί σε σχέση με τη δεκαετία του 60. Είναι πέντε φορές ε, μεγαλύτερη ε, τώρα από ότι στη δεκαετία του Και η μετάβαση από τη, τα, τις παραδοσιακές ε, διατροφικές συνήθειες στις αναπτυσσόμενες χώρες προς ε, τη, τα επεξεργασμένα τρόφιμα έχουν, έχει οδηγήσει σε μεγάλη εξάρτηση από τις εισαγωγές στον τομέα των τροφίμων. Και το θέμα που τίθεται είναι πώς μπορούμε να διαφρόσουμε τις προτεραιότητές μας, διότι <clears throat> τις τελευταίες δύο-τρεις δεκαετίες η κατάσταση έχει αλλάξει προς το χειρότερο. Παράδειγμα, η μετάβαση στην μεγαλύτερη ε, παραγωγή κρέατος για κάθε κιλό ζωικής πρωτεΐνης απαιτεί 5 κιλά φυτικής πρωτεΐνης. 5 φορές μεγαλύτερο όγκο δηλαδή. Απαιτείται επίσης ε, πολύ μεγαλύτερο όγκος νερού. Χρειάζεται λοιπόν να αλλάξουμε τις προτεραιότητές μας. Βρεθήκαμε στην ε, Γένοβα κατά την ε, διάσκεψη για το διεθνές εμπόριο και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή στον τομέα του διεθνούς εμπορίου είναι το εμπόριο τροφίμων. Θα είναι λοιπόν και αυτό ένα από τα πολύ ευαίσθητα ζητήματα και θα πρέπει να αποφύγουμε τον ε, ανταγωνισμό ανάμεσα στην παραγωγή τροφίμων και στην παραγωγή βιοκαυσίμων, διότι και αυτό επιδίνωσε την κατάσταση στα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με δήλωση του κ. Λίψκη στο ε, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε μια ακρόαση που έγινε στο ε, Κογκρέσο των Ηνωμένων ο κ. Λίψκη είπε ότι το μερίδιο των βιοκαυσίμων ε, στην διαμόρφωση ε, των τιμών τροφίμων ε, το μερίδιο ανέρχεται σε 70%, στην περίπτωση της σόγιας ανέρχεται σε 40%. θα έπρεπε να τριπλασιάσουμε το, την επιφάνεια της ε, αρρώσιμης γης για να παράγουμε ε, τρόφιμα για όλον τον πλανήτη, εάν συνεχίζαμε αυτό το σύστημα. Χρειάζεται λοιπόν να αλλάξουμε προτεραιότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ προσωπικά. Βρίσκω πολύ σημαντική τη γνωμοδότηση αυτή. Θέλαμε λοιπόν να γνωμοδοτήσουμε στην Επιτροπή Άγκρη για το θέμα αυτό, Γεωργία και Διεθνές Εμπόριο, διότι όπως ε, γνωρίζετε η Γεωργία είναι ίσως ο πιο ευαίσθητος τομέας στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και ε, η δεσπόσα θέση στον ε, τομέα της Γεωργίας είναι προ... προτεξιονιστική, μη σας πω αντιεμπορική τα γεωργικά συμφέροντα φυσικά θα πρέπει να λαμβάνονται απόψη και θα πρέπει να προστατευτούν τα νόμιμα συμφέροντά τους. Εμείς όμως ως μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου θα πρέπει να έχουμε μία συνολική και ισορροπημένη εικόνα του εμπορίου, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας να λαμβάνουμε υπόψη δηλαδή και τις επιχειρήσεις ε, και τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές. Πιστεύω λοιπόν ότι πρόκειται για εξαιρετική ευκαιρία για μας να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Και είμαι βέβαιος ότι η συγγήτριά μας θα μπορέσει να υποβάλει μια ισορροπημένη και σωστή γνωμοδότηση. Δίνω το λόγο στον κύριο Ζαντώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, το είπατε, είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση και είναι ουσιαστικό η Επιτροπή να εξετάσει σοβαρά το θέμα. Η Ευρώπη έχει γίνει ο πρώτος εισαγωγέας ακατέργαστων των γεωργικών προϊόντων πριν από την Κίνα το μισό των εισαγωγών της είναι φυτικές πρωτεΐνες για την τροφή των κοπαδιών στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να το συνδέσουμε αυτό με την μελλοντική μεταρρύθμιση της ΚΑΠ πρέπει η συμφωνία του Blair House να καταργηθεί. Δεν έχει κανένα νόημα πλέον εφίσταται αυτή η συμφωνία. Δηλαδή είναι καταχρηστική πλέον αυτή η συμφωνία που ρυθμίζει ε, τους, ε, ε, τις, ε, ε, την εισαγωγή ολικών πρωτεϊνών. και των ζωοτροφών γιατί έχει ξεπεραστεί εντελώς αυτή η αντίληψη για το πώς εκτρέφονται ζώα στην Ευρώπη. Στην ε, Γαλλική Προεδρία θα βρίσκεται και το θέμα και στην, ε, στους ε, G20 δηλαδή για την τροφιμική για τις τροφ φημικές κερδοσκοπίες στις διεθνείς αγορές. Δηλαδή, ορισμένα τρόφιμα χρησιμοποιούνται ως αντικείμενα κερδοσκοπίας. Πρέπει λοιπόν να βρεθούν μέτρα που να εμποδίζουν την κερδοσκοπία των γεωργικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Τώρα, διεθνείς συμφωνίες όλες οι συμφωνίες που κάνουμε Όλες οι συμφωνίες που κάνουμε πρέπει να έχουν κατά νου το θέμα της μετατόπισης των γεωργικών επιχειρήσεων. Ο μεγαλύτερος εκτροφέας πουλερικών βρίσκεται στη Γαλλία. Λέγεται ντου. Λοιπόν, παράγει τεράστιες ποσότητες, ε, εκτρέφει τεράστιες ποσότητες κοτόπουλο στη Γαλλία, αλλά η έδρα του είναι στη Βραζιλία. Οπότε όταν βρίσκεται στη Βραζιλία τι κάνει, διαπραγματεύεται τις ε, διευκολύνσεις και την απολευθέρωση των εισαγωγών από τη Βραζιλία. Πρέπει λοιπόν η Κομισιόν να έχει την δυνατότητα να διερευνήσει περισσότερο αυτές τις επιχειρήσεις, ε, τι διαχειρίζονται, πόσες επιδοτήσεις παίρνουν ε, και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένε Πολιτείες ε, οι οποίοι διαφορούν πλήρως για το πού παράγεται η τροφή. Απλώς εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι να ταξιδεύει αυτή η τροφή. Επίσης, πρέπει να δούμε και τις επιπτώσεις στις εξαγωγές. Εμείς διαπιστώσαμε ότι ορισμένες επιδοτήσεις πέρασαν από το πράσινο στο μπλε ή στο κίτρινο κουτί. Λοιπόν, το dumping στις διεθνείς αγορές ε, έβαλε σε κρίση πολλές, ε, ε, πολλές παραγωγές, κυρίως στο νότο της Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσει αυτό και το προϊόν όταν, πουλείται, να, όταν πουλιέται να αντικατοπτρίζει τις πραγματικές του τιμές και την κοινωνική τιμή, περιβαλλοντικό κόστος και κόστος παραγωγής. Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως το υπογραμμίσατε κι εσείς και πολλά μέλη της Επιτροπής σας, η έκθεση αυτή είναι πολύ σημαντική και η ευκαιρία είναι καταπληκτική για να μιλήσουμε για το εμπόριο στα τρόφιμα. Το εμπόριο αποτελεί ένα παράγοντα το οποίο, ο οποίος ε, προωθεί ιδιαίτερα την οικονομική ανάπτυξη και το εμπόριο στα τρόφιμα έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Το γεωργικό αυτό εμπόριο μεταξύ του 2000 και του 2009 διπλασιάστηκε σε παγκόσμιο επίπεδο. Είδαμε ότι έχουν αυξηθεί οι εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ Νότου και Νότου με πολύ μεγάλη αύξηση στα έσοδα, τα κέρδη, ιδίως στην Ασία. Αλλά όπως είπαν και ορισμένοι, υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις οι οποίες οργανώνουν πλέον την παραγωγή τους σε παγκόσμιο επίπεδο σε επίπεδο παγκόσμιας αλυσίδας εμπορικών συναλλαγών. Η παγκόσμια βέβαια οικονομική κρίση επηρέασε πολύ το εμπόριο στα τρόφιμα. Αν συγκρίνουμε όμως το εμπόριο σε γεωργικά προϊόντα με το συνολικό εμπόριο υπηρεσιών που μειώθηκε το 2009 κατά 12%, το εμπόριο στα τρόφιμα μειώθηκε μόνο κατά 3%. Είχαμε βέβαια μια πολύ σημαντική μείωση σε επίπεδο αξίας, ακριβώς επειδή μειώθηκε πάρα πολύ η τιμή των γεωργικών προϊόντων σε σχέση με το 2008. Θα ήθελα να σας δώσω τώρα κάποια δεδομένα προκειμένου να είμαστε θέση να δούμε ποια είναι η θέση που κατέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τους υπόλοιπους εταίρους μας όσον αφορά το εμπόριο σε γεωργικά προϊόντα και ενδεχομένως τα αριθμητικά αυτά δεδομένα να σας ενδιαφέρουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι Συγγνώμη, οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι ο σημαντικότερο εμπορικό μα εταίρο και μαζί με τι Ηνωμένε Πολιτείε είμαστε και εμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από του μεγαλύτερου εξαγωγεί ε, προϊόντων. Το 2009 104 δισεκατομμύρια δολάρια ήταν η αξία των προϊόντων που εξάγαμε. Και έχουμε ένα μερίδιο τη αγοράς εξαγωγών που βρίσκεται μόλις κάτω από το 18%. Η Βραζιλία είναι η τρίτη μεγάλη δύναμη. 14 δισεκατομμύρια είναι η αξία των εξαγωγών της Βραζιλίας από το 1999 στο 2001 και πέρασε στα 55 δισεκατομμύρια το 2009. Και ουσιαστικά έχει ξεπεράσει τον Καναδά που είχε κατήχε την τρίτη θέση παλιότερα. Όσον αφορά τις αγωγές, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας στον κόσμο. Οι εισαγωγέ μας το 2009 φτάσανε τα 107 δισεκατομμύρια δολάρια. Είμαστε οι πρώτοι και στη συνέχεια ακολουθούν με 77 οι Ηνωμένε Πολιτείε με 77 δισεκατομμύρια. Η Ιαπωνία και η Κίνα η Κίνα πρόσφατα μπήκε στην ομάδα αυτή των μεγάλων εισαγωγών, βρίσκονται στην τρίτη και την τέταρτη θέση αντίστοιχα. Οι εισαγωγές της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν το 19% των παγκοσμίων εισαγωγών σε ε, προϊόντα όσον αφορά την γεωργία πάντα. Να πω τώρα κάποια λόγια, κάποια λόγια για την δομή των εξαγωγών μας, τη διάρθρωσή τους. Τα βασικότερα προϊόντα τα οποία εξάγουμε Πρόεδρος, είναι απλώς η πρώτη ανταλλαγή απόψεων που μπορείτε να συντομεύσετε την παρέμβασή σας. Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πολύ καλά. Ήθελα απλώς να σας δείξω ότι οι βασικές μας εξαγωγές είναι τελικά προϊόντα, τα οποία τις περισσότερες φορές πηγαίνουν προς χώρες και πλούσιους καταναλωτές. Αναφέρομαι τελικά προϊόντα της ποιότητος. Και οι εισαγωγές μας είναι κυρίως εισαγωγές από αναπτυσσόμενες χώρες και ουσιαστικά είναι ζωοτροφές και εισάγουμε και πολλά τροπικά προϊόντα όπως καφέ, κακάο και μπανάνες. Αν δούμε λοιπόν την δομή του διεθνού μας εμπορίου, βλέπουμε ότι η μεγάλη μας δύναμη είναι η πολύ υψηλή ποιότητα και προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας. Προκειμένου όμω να διατηρήσουμε την ποιότητα αυτή χρειαζόμαστε και τι απαραίτητες εισαγωγέ για να είμαστε θέσει να παράγουμε στη συνέχεια τα προϊόντα αυτά υψή τη ποιότητος. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η ποιότητα και η υψηλή προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας αποτελούν το μεγάλο πλεονέκτημα που έχουμε στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου και θα αποτελούν το μεγάλο πλεονέκτημα που θα έχουμε στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου. Επίσης, η πολύ ευφυής προώθηση των προϊόντων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης και η στάση μας όσον αφορά τις διεθνείς διαπραγματεύσεις, καθώς επίσης και η προστασία συγκεκριμένων προϊόντων, ιδίως όσον αφορά τη γεωγραφική ένδειξη, αποτελούν τα βασικά κριτήρια τα οποία θα πρέπει να διαμορφώνουν την πολιτική μας και στο μέλλον. Είμαι στη διαθεσή σας για οποιασδήποτε πληροφορίες χρειάζεστε για την έκθεσή σας οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιο συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση γεωργίε στη διάθεσή σα για να συμβάλλουν για τη σημαντική αυτή έκθεση. Σα ευχαριστώ. Στο μέλλον θα έχουμε άλλε ευκαιρίε ανταλλαγή απόψεων και θα είναι πολύ χρήσιμε οι θέσεις σα για τη γνωμοδότησή Μα. Υπάρχουν ε, άλλε παρατηρήσει. Η συγκήτρια έχει τελικέ παρατηρήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσου ε, συμμετείχαν στη συζήτηση αυτή. Μία παρατήρηση. Οι φτωχότερε ε, ε, χώρες του κόσμου ε, ηγούνται από δικτάτορες της αριστεράς. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να ε, κονίσουμε μια έκθεση η οποία να αντικατοπτρίζει τη βασική θέση της Επιτροπής μας. Δυστυχώς η έκθεση αυτή δεν θα μπορέσει να αλλάξει τον κόσμο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Δύο πράγματα. Εγώ άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το οποίο είπε η κυρία. Αλλά δεν ξέρω γιατί από πού το έβγαλε δηλαδή ότι όλες οι αναπτυσσόμενες χώρες κυβερνώνται από δικτάτορες της αριστεράς και γιατί όχι δικτάτορες της δεξιάς. Λοιπόν και στο κάτω-κάτω είναι αποδεδειγμένο πλέον ότι ήταν και δικτάτορες της δεξιάς μέχρι και φασίστες από, και κατά καιρούς τους οποίους υποστηρίξατε. Μπορούμε να το συζητήσουμε και εκτός Επιτροπής αυτό. Το σχέδιο έκθεσης προβλέπεται για τις 25-26 Οκτωβρίου και ας προχωρήσουμε τώρα σύντομα στο σημείο 13 χορήγηση εγγύησης Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις για σχέδια εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγγητής μας είναι ο William Dartmouth. του EFT. Όπως ξέρετε υπήρξε ενδιάμεση αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και η Κομισιόν προτείνει να συνεχιστεί, να συνεχιστεί και να επεκταθεί η ε, εγγύηση προς την τράπεζα. Σας παρακαλώ, δείξτε λίγο σεβασμό. I will give the floor to να δώσω το λόγο στο William Dartmouth. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι ένα από τα προνόμια της Επιτροπής μας ε, είναι η εξαιρετική προεδρία σας ε, το τελευταίο χρόνο και ζητώ συγγνώμη που, που ε, μου διέφυγε το γεγονός ότι ένα θέμα της μέσης διάταξης είχε μεταφερθεί σε άλλο σημείο. Παρ' όλα αυτά οι παρατηρήσεις μου ισχύουν και σκέφτομαι να τις βάλω και στην ιστοσελίδα μου. Όσον αφορά το ότι οι εκθέσει μπορεί να μην αλλάξουν τον κόσμο, σίγουρα μπορούμε να προσπαθήσουμε και θα συμφωνούσα με του συναδέλφου μου εδώ στα αριστερά μου. Θα περιοριστώ σε μια πολύ σύντομη παρουσίαση. Ε, χάρη στην πολύ καλή δουλειά της γραμματείας γνωρίζω πολύ περισσότερο για το θέμα από ό,τι πριν, γνώριζα πριν 24 ώρες. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπάρχει για να... Μια σύντομη παρουσίαση θα ε, για να στηρίξει και παραθέτω ε, καλές επενδύσεις οι οποίες να προωθούν τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ε, οι στόχοι όσον αφορά το δανεισμό σε περιοχές ε, που να μην καλύπτει η πρόταση οι τράπεζα έχουν να κάνουν με ε, την προνταξιακή βοήθεια, την ε, φόρο ενέργεια, την στήριξη της παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Ε, ιδιαίτερα στηρίζω τη ρήτρα στο άρθρο 5 που λέγει ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα διαβολεύεται την, την υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρότι λοιπόν πρόκειται για τράπεζα και είναι τράπεζα, δηλαδή τονίζει χρήματα, πρόκειται και για έναν φορέα που στόχο έχει να προωθήσει την ατζέντα της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής. Τώρα προτείνεται και γι' αυτό το θέμα αυτό έχει υποβληθεί στην Επιτροπή μας. Ε, προτείνεται το επίπεδο των ευρωπαϊκών επενδύσεων που ανέρχεται σε 24,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι εγγυήσει αυτές ουσιαστικά ισοδυναμούν με ε, ε, κρυφά περιουσιακά στοιχεία και όλα αυτά στηρίζουν 500 δισεκατομμύρια ε, ευρώ ε, δυνατότητας δυναμισμού και, ε, δανεισμού και 5% εγγυήσεις είναι αρκετά υψηλό ποσοστό. Προτείνεται λοιπόν να δοθούν άλλα 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε εγγυήσεις, να φτάσουμε στα 77,8 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων τα 2 δισεκατομμύρια θα καταμεθούν ιδιαίτερα για να καταπολεμηθεί η ε, αλλαγή του κλίματος. Για την καταπολέμηση, όχι για να επιφέρει περισσότερη, μεγαλύτερη αλλαγή του κλίματος. Θα ήθελα επίσης να πω ότι υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες όσον αφορά κάποιες χώρες και είναι κάπως τυχαίες. Οι πέντε χώρες στις οποίες θα δοθεί προτεραιότητα είναι η Ισλανδία για προενταξιακή ε, βοήθεια, η Λευκορωσία για την ιδιωτικοποίηση, η Λιβύη για μέτρα αντιμεταναστευτικά και κατά του AIDS, το Ιράκ για την υποδομή και η ε, Καμπότζια για ε, την ε, για την ανάκαμψη της χώρας. Ε, αυτά προς στιγμή και περιμένω να ακούσω τις ε, παρατηρήσεις της Επιτροπής σας. Ε, πολύ αργότερα θα σας υποβάλω και τη δική μου γνώμη. Πρώτον, να δώσω το λόγο στους άλλους βουλευτές να πω ότι η δεύτερη ανταλλαγή απόψεων θα γίνει στις 30 Αυγούστου και η εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης 28 ή 29 Σεπτεμβρίου. Ο κύριος Ζαντώ que η ΕΤΕ είναι πολύ καλό πράγμα να έχει μία εντολή για την αλλαγή του κλίματος. Είναι πολύ καλό πράγμα. Διότι οι επενδύσεις ε, του, σχεδίου, του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάκαμψης ε, αν προσανατολίζεται για την ε, οικολογική ανάπτυξη κλπ. είναι πολύ καλό πράγμα. Τώρα, το να αυξηθεί δύο δις αυτή η εντολή για το κλίμα τότε θέλουμε να ξέρουμε πολύ, πολλά περισσότερα. Δηλαδή ποιες είναι οι δυνατότητες της ΕΤΕ να διευρύνει την εντολή, να επεκτείνει την εντολή την οποία έχει στον τομέα αυτό και τι σχέδια υποβάλλονται. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πολλές, πολλές φορές ε, είπε ότι δεν πρέπει να υποστηρίζει ε, στις ε, να υποστηρίζει η ΕΤΕ επενδύσεις για ορυκτά ορυκτές πηγές ενέργειας αλλά να ε, προσπαθεί να ε, προσανατολιστεί προς άλλα σχέδια, φράγματα ή οτιδήποτε άλλο. Ε, να, μάλλον να αποκλείει τα φράγματα ε, τους, τις θερμοηλεκτρικές ε, εγκαταστάσεις, ε, την εκμετάλλευση πετρελαίου και άλλων ορυκτών ε, πηγών ενέργειας. Ο Σκιώδης ηγητής από το ΕΛΚΑ, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται σαφώς για μια πρώτη απλώς ανταλλαγή απόψεων, θα είμαι λοιπόν σύντομος. Θα ήθελα καταρχάς να χαιρετήσω το γεγονός ότι γίνεται αυτή η ενδιάμεση αναθεώρηση Βρισκόμαστε στο μέσο των δημοσιονομικών προοπτικών 2007-2013 και θα ήθελα να τονίσω κάποια νέα στοιχεία όσον αφορά την εντολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Την αντικατάσταση του περιφερειακού στόχου από τους οριζόντιους στόχους. Προφανώ θα μπορούσαμε να μιλήσουμε περισσότερο για του στόχου και για το πώ καταρτίζονται ή θα μπορούσαμε να συζητήσουμε αν θέλετε αν είναι ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη Επιτροπή μα να απαγορεύσει κάποιου ε, στόχου. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε καλύτερα να θέτουμε τα κριτήρια για την κατάρτιση των στόχων. Αυτό να συζητάμε. Ως βουλευτή προερχόμενο από μια χώρα που είναι από τα πιο νέα μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελα να τονίσω το ότι ε, στόχοι όπως ε, η περιβαλλοντική υποδομή, η ανάπτυξη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένας πολύ σημαντικός στόχος για το ΕΛΚ βέβαια, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι στόχοι λοιπόν αυτοί είναι πολύ σημαντικοί και ορίζονται πολύ καλά. Όσον αφορά τώρα τα νέα στοιχεία της εντολής Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, και όσον αφορά πιο συγκεκριμένα την ιδέα του περιφερειακού ορισμού των ε, προτεραιοτήτων, θα πρέπει οι ε, χώρες ε, της πολιτικής γειτονίας και οι χώρες που βρίσκονται σε προενταξιακό στάδιο να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της δραστηριότητας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Οι Ευρωπαϊκές Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης και οι Ευρωπαϊκές Προενταξιακές Συμφωνίες είναι πολύ σημαντικές και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να χρηματοδοτούνται περισσότερο, τουλάχιστον να αποτελούν προτεραιότητα των δραστηριοτήτων και των επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Σας ευχαριστώ. Thank uh, Σας ευχαριστούμε. George ε, Κούτας, σκιώδης συγητής ε, από τους σοσιαλιστές. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι τα νέα στοιχεία που έχουμε στην Συμφωνία για τη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι στοιχεία ιδιαίτερα θετικά. Μπορούμε να καθοδηγήσουμε πλέον την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προς, τις, τα προγράμματα εκείνα τα οποία θα στοχεύουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τις αηφόρες μεταφορές, την κοινωνική και οικονομική υποδομή και ανάπτυξη. Είναι πολύ σημαντικό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Κατά αυτόν τον τρόπο θα τονωθεί η οικονομία και θα καταπολεμήσουμε την ανεργία. Είναι σημαντικό επίσης να μπορούμε να εγγυηθούμε τη βιώσιμη ανάπτυξη των εταίρων μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στα πλαίσια Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε ευνοϊκές συνθήκες για το εμπόριο το ποσό των δανείων που δίνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιστοιχεί στο ίμιση των δανείων που εκχωρούνται από την Παγκόσμια Τράπεζα. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί πλέον ένα πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό μηχανισμό που μπορεί να μας επιτρέψει να πετύχουμε τους στόχους συνεργασίας που έχουμε με τις χώρες εταίρους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν κατακλείδη θα ήθελα να σας πω ότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να έχουμε ετήσιες αξιολογήσεις τη αποτελεσματικότητας των δανείων, προκειμένου να έχουμε ένα υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας για τη χρήση των δανείων και προκειμένου να καταφέρουμε να μειώσουμε το γραφειοκρατικό άχθος. Ευχαριστώ. Μου λένε ότι βρίσκεται εδώ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θα χαρώ λοιπόν να δώσω το λόγο στον κύριο Αλεσάνδρο Καράνο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 για τις εγγυήσεις ε, μετά από την ε, νέα ε, απόφαση του δικαστηρίου. Επικροτούμε την εξέλιξη αυτή και επικροτούμε και τη συμμετοχή της Επιτροπής ΣΥΝΤΕ καθώς και το σημαντικό ενδιαφέρον που δείχνεται για τις εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως που όπως είπατε ότι αυξάνονται σταθερά τα τελευταία χρόνια μέχρι που φτάσαμε στο ε, ε, παρόν επίπεδο χρηματοδότησης ε, που ανέρχεται στο ύψος του, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Περιφερειακής Ανάπτυξης και περίπου στο, μισό της Παγκόσμιας Τράπεζας. Γνωρίζετε την ενδιάμεση αναθεώρηση. Ξέρετε ότι και η ΕΚΟΦΗΝ έχει αναφέρει τις βασικές της προθέσεις όσον αφορά την πρόταση αυτή. Θα θέλαμε να τονίσουμε την ανάγκη να ευθυγραμμίσουμε τις φιλοδοξίες μας με τις απαιτήσει της εντολής. Ε, αυτό σύντομα αναφέρθηκε. Υπάρχει ανάγκη να ευθυγραμμιστούν προσεκτικά όλες αυτές οι πτυχές, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για την ανάπτυξη των ε, ε, δραστηριοτήτων του, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάπτυξη. Αυτό απαιτεί ιδιαίτερη μια συγκεκριμένη προσέγγιση και γνωρίζετε ότι στηρίζουμε τις ε, πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, πολιτικά λογοδοτούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πολύ ευχαρίστω ε, θα διευκρινίσουμε οποιοδήποτε στοιχείο της πρότασης αυτής μαζί με τους συναδέλφους από την Επιτροπή μας. Περιμένουμε να λάβουμε την καθοδήγησή σας για συγκεκριμένα ζητήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Ράμστορ. Σύντομη παρατήρηση παρακαλώ, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Τελειώνει ο χρόνος. Ναι. Σας έδωσα το λόγο. Παρακαλώ απλά να είσαστε σύντομος. Ε, σύντομα, έχω δύο παρατηρήσεις. Ε, καταρχήν, στο κείμενο αναφέρεται το πρόβλημα ε, της ε, παροχής συμβουλών από ε, της διαβούλευσης με, τις, με την Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων. Αλλά θα πρέπει να συμμετέχουμε και εμείς για να συμπληρώσουμε το κενό που υπάρχει, διότι είναι πολύ σημαντικό να αποφύγουμε κάποιους κινδύνους στον τομέα αυτό για το μέλλον. Και η δεύτερη παρατήρηση να δώσω συνέχεια στην επιχειρηματολογία του κυρίου Βίνκλερ. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε ζητήματα, σε πράγματα εφικτά. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ένταξη των Βαλκανίων, διότι χωρίς τα Βαλκάνια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι ποτέ πλήρης. Ε, η Κομισιόν έχει παρατηρήσεις καθότι συζητάμε πρόταση της Κομισιόν. Στέφαν Άπελ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε πολύ σύντομα κάποιες παρατηρήσεις. Η πρόταση αυτή ακολουθεί απέτηση σε απόφαση της, ε, του Συμβουλίου να ε, υποβάλλεται ενδιάμεση αναθεώρηση. Η πρόταση που έχει υποβληθεί τώρα από την Κομισιόν προτείνει διάθεση των ε, επιπλέον 2 εκατομμυρίων για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Και θέλουμε επίσης να έχουμε περισσότερες επιλέξιμες χώρες, ε, να προσταθούν δηλαδή αυτές που, αναφέρονται στο κείμενο. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι η ε, μεροντική χρηματοδότηση θα περιοριστεί στις χώρες αυτές. Μιλάμε για ε, διεύρυνση της χρηματοδότησής μας που θα καλύπτει και αυτές τις χώρες. Σημειώσαμε ότι το Συμβούλιο έχει οθετήσει μια θετική ε, γενική προσέγγιση και γι' αυτό προσβλέπουμε σε ε, ομαλή ε, εκτέλεση των σχεδίων μας με την γρήγορη υιοθέτηση. Ο κύριος Ντάρθμουθ, να σας πω ότι ε, μόνο εδώ όταν μιλάω μου ζητάνε να ανάψω το μικρόφωνο. Σημείωσα τις παρατηρήσεις των ε, συναδέρφων. Μείνετε ήσυχοι. Ε, σίγουρα θα ασχοληθούμε με το πού θα δοθούν τα χρήματα για την καταπολέμηση του κλίματος. Ο κύριος Βίνκλερ πολύ σωστά είπε αυτό που δεν είπα εγώ, ότι η χρηματοδότηση τώρα πια θα είναι οριζόντια και όχι περιφερειακή, το οποίο διορθώνει αυτό που είπε ο κύριος, ε, το οποίο αντίκειται σε αυτό που είπε ο κύριος Άντροφ για τα Βαλκάνια. Επίσης με ενδιέφερε το άλλο που αναφέρθηκε, ε, ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανέρχεται στο μισό περίπου τη Παγκόσμια Τράπεζα όσον αφορά το δανεισμό και ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Περιφερειακής Ανάπτυξη ε, είναι περίπου ε, εξίσου μεγάλη, το οποίο σημαίνει ότι ε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Περιφερειακής Ανάπτυξης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, δανείζουν περίπου όσα χρήματα δανείζει η Παγκόσμια Τράπεζα. Προσλέπω στην περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων και τις περαιτέρω παρατηρήσεις σας να ευχαριστήσω και τους δύο εκπροσώπους της Κομισιόν για τις πολύ χρήσιμες και επίκαιρες παρατηρήσεις τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να ζητήσω συγγνώμη στον ε, προσκεκλημένο μας ε, τον ε, πρέσβη της Νοτιού Αφρικής για την καθυστέρηση αλλά θα πρέπει να κλείσουμε τα άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη πρωτού τον ακούσουμε. Παρακαλώ λοιπόν να είναι υπομονετικός. πιστεύω ότι αυτό θα είναι ε, σύντομο θέμα στη ημερήσια διάταξη. Έχουμε το 14 πίσω του κανονισμού ε, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο Γενικό Προπολογισμό των ε, Ευρωπαϊκών ε, Κοινοτήτων όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Μιλάμε δηλαδή για τη χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Η συγητή μα είναι ο Κάντερ Αρίφ από του Σοσιαλδημοκράτε και του δίνω το λόγο. Παρακαλώ. Merci rapidement. Euh, σας ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Κάποιες διευκρινήσεις θέλω να δώσω για το χρονοδιάγραμμα εργασίας για το ζήτημα αυτό. Όπως το γνωρίζετε, μια γενική συμφωνία στις 21 Ιουνίου είχαμε για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Την προηγούμενη εβδομάδα στην Επιτροπή ΑΘΕΤ και στη συνέχεια στην Ολομέλεια ψηφίσαμε για την σύσταση της νέας αυτής υπηρεσίας νέα υπηρεσία η οποία θα έχει έναν κεντρικό κανονισμό και δύο επιπλέον κανονισμούς, έναν δημοσιονομικό και έναν υπηρεσιακό κανονισμό. Εγώ εργάστηκα για τον δημοσιονομικό κανονισμό. Πολλές φορές τα πράγματα εμφανίζονται κάπως πολύπλοκα. Επομένως θα ήθελα να πω ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα έχει ένα προπολογισμό λειτουργίας. Όλες οι αντιπροσωπείες υπάγονται στην υπηρεσία αυτή. Υπάρχει ένας προϋπολογισμός που δίδεται από τον δημοσιονομικό κανονισμό και η γνωμοδότηση επί της οποίας εγώ εργάζομαι λέει κάτι σημαντικό για την Επιτροπή μας. Στην περίπτωση διαφοράς, στη χρήση του προπολογισμού και συγκεκριμένα όταν αυτό έχει να κάνει με την πολιτική για το εμπόριο, η διαφορά αυτή θα πρέπει να διευθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι από την ΥΠΑ το εκπρόσωπο. Δηλαδή, σε περίπτωση διαφοράς, σε περίπτωση διένεξης, οποιοδήποτε εταίρος μας από τρίτη χώρα θα μπορεί να απευθυνθεί βέβαια είτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε στην ύπατη εκπρόσωπο, αλλά την τελική απόφαση για την επίλυση της διαφοράς θα τη λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό γιατί το διεθνές εμπόριο αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι της ΥΠΑΤΗ εκπροσώπου. Ελπίζω να διευκρίνησα τα πράγματα για το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ. Πρόκειται λοιπόν για μια έκθεση με αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή την Επιτροπή Προπολογισμού. Προθεσμία καταβολής ε, τροπολογιών είναι η 16η Ιουλίου. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας για τη γνωμοδότηση αυτή στις 30 Αυγούστου. Δεν έχουμε ορίσει ακόμα τους σκιώδεις ηλιτές Πέρα από τον κύριο Ζαλέσκι από το ΕΛΚ υπάρχουν ε, άλλα μέλη της Επιτροπής που θέλουν να πάρουν τώρα το λόγο. Όχι. Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν. Μπράντον Κούγκαν ονομάζομαι κύριε Πρόεδρε και θα μιλήσω εξ ονόματο της κυρίας Γκίλγκερστ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήμουνα και χθε στην Επιτροπή σας, αυτή είναι η δεύτερη μου μέρα και θέλουμε να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να συσταθεί και να λειτουργήσει αυτή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης με ένα πολύ καλό σύστημα δημοσιονομικής διαχείρισης και θέλουμε να μπορέσει να ξεκινήσει τις λειτουργίες της το συντομότερο δυνατό, γιατί έχει πολύ μεγάλη πολιτική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η υπηρεσία. Άκουσα τα σχόλια του εισηγητή. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η έκθεση αυτή, πώς θα ψηφίσετε για την έκθεση αυτή, για την πρότασή σας στην Επιτροπή. Ουσιαστικά είμαστε θετικά διακείμενοι για τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα και όπως αναφέρεται ήταν πολύ σημαντική και έκφαση του τετραμελούς διαλόγου που έλαβε χώρα στη Μαδρίτη και που ήταν ουσιαστικά μια έκφαση καθοριστική για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε. Συντάξει γνωμοδότης ήταν ο κύριος Καντέρ Αρίφ. Θέλετε κύριε Αρίφ το λόγο πρωτού κλείσουμε το ζήτημα αυτό. Μην ξεχνάτε ότι έχετε δύο μέρες για να υποβάλλετε τροπολογίες. 16 Ιουλίου είναι η προθεσμία στις 12 το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Περνάμε τώρα στο σημείο 15. Ανταλλαγή απόψεων με τον πρέσβη της Νοτιοαφρικής, τον κύριο Ανίλα Σούκλαλ. Καλώς ήρθατε κύριε Σούκλαλ στην Επιτροπή μας. Έχουμε συναντηθεί και στο παρελθόν προσωπικά Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε εδώ μαζί μας σήμερα και που θα έχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε στην Επιτροπή μας. Όπως γνωρίζετε, η Νότιος Αφρική είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός μας εταίρος στην Ήπειρο της Αφρικής. Οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση διεξάγονται από την συμφωνία FTA μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νοτιοαφρικής. Η Νότιος Αφρική ανήκει επίσης και στην ΣΑΔΚ, δηλαδή την ε, ε, κοινότητα ανάπτυξης του εμπορίου στην ε, Νότιο Αφρική, στην Μεσημβρινή Αφρική. Τον Οκτώβριο οργανώσαμε μία αντιπροσωπεία η οποία θα επισκεφθεί την Νότιο Αφρική σε συνεργασία με τις αρχές της Αφρικής και με τις κοινοβουλευτικές αρχές της χώρας αυτής. Νομίζω ότι η επίσκεψη αυτή θα είναι πολύ χρήσιμη και θα επιτρέψει στην Επιτροπή μας να καταλάβει καλύτερα πώς λειτουργεί αυτή η ταχαίως αναπτυσσόμενη οικονομία της Αφρικής θα καταφέρουμε να καταλάβουμε επίσης καλύτερα τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Νότιος Αφρική στις ε, εμπορικές διαπραγματεύσεις της παγκόσμιας που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω επίσημα τον πρέσβη της Νοτιοαφρικής κύριο, κύριο Άνιλ Σούκλαλ και θα ήθελα επίσης να σας συγχαρώ και εσάς και του συνεργάτες σας για την καταπληκτική διοργάνωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι πραγματικά μπορεί να είστε περήφανοι για τη χώρα σας και όλοι οι Νοτιοαφρικάνοι μπορεί να είναι περήφανοι για την διεξαγωγή της, του πρωταθλήματος. έδειξε η Αφρική ότι είναι σε θέση να οργανώνει καταπληκτικά εκδηλώσεις παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Είστε κύριε Σούκλαλ, πρέσβης της Νοτιοαφρικής ε, στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και έχετε το λόγο. Uh, uh, ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου καταρχήν να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας προς την προς εσάς και την ε, Επιτροπή σας ε, που μπορέσαμε να ε, βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Σας ευχαριστούμε και για τα συγχαρητήρια σας για την οργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Χαιρόμαστε που το Κύπελο κατέληξε σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση κερδίζει το Κύπελο σε περίπτωση διοργάνωσης του πρωταθλήματος εκτός. Πολύ σύντομα θα καλύψω τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτού προχωρήσω σε θέματα διανοητικής διευθυνσίας κλπ. Όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι για μας στρατηγικός εταίρος, είναι η περιφέρεια που Σύντομα μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 1994 ε, ήταν μία από τις ε, πρώτες περιφέρειες ε, που ήρθαν σε επαφή μαζί μας. Ήταν η πρώτη περιφέρεια που ήρθε σε επαφή μαζί μας. Ξεκινήσαμε λοιπόν τις διαπραγματεύσεις και ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις το 1999 και τέθηκαν σε ισχύ 1η Ιανουαρίου του 2000. Το TCA καλύπτει τέσσερις τομείς, πολιτικό διάλογο, εμπόριο και την ε, σύναψη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου, αναπτυξιακή συνεργασία και επίσης ε, οικονομική συνεργασία πρόκειται για ε, σημαντική συμφωνία, νομικά δεσμευτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το και την όθιο Αφρική. μέχρι το 2005 λειτουργούσε πολύ καλά. Τότε θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επεκτείνει την ε, συμφωνία αυτή και στον ε, πρόεδρό μας, τον κύριο Μπέκη, υποβλήθηκε ε, ανεπίσημο έγγραφο που είχε να κάνει με την επέκταση της στρατηγικής συνεργασίας. Στον διάλογο ε, που ε, ονομάστηκε από το κίτρινο δέντρο που είναι το εθνικό δέντρο της Νοτιού Αφρικής ε, κόμπα κόμπα που ίσως να ξέρετε ότι στην παράδοση της Νοτιού Αφρικής οι συμφωνίες συνάπτονται κάτω από ένα τέτοιο δέντρο. Ε, αυτή λοιπόν είναι η συμφωνία η οποία ισχύει αυτή τη στιγμή και διέπει τις ε, σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νοτιού Αφρικής. Ε, γίνεται κάθε χρόνο διάσκεψη κορυφής. φέτος η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διοργανώσει τη συνάντηση αυτή εδώ στις Βρυξέλλες στις 28 Σεπτεμβρίου όπου θα συμμετάσχει και ο Πρόεδρός μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από ο σημαντικότερο εμπορικό μα εταίρο, είναι και η μεγαλύτερη πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων ε, τουρισμού. Το είδαμε αυτό τώρα και με το παγκόσμιο κύπελο. Μεγάλος αριθμός ε, ε, ποδοσφαιρόφιλων έφτασαν στην Νότια Αφρική και φυσικά είναι και ο μεγαλύτερος εταίρος μας όσον αφορά την αναψυχική συνεργασία. για το διάστημα 2007-2013 δόθηκαν ε, στην ε, Νότια Αφρική 980 εκατομμύρια ευρώ και άλλα 900 από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μέχρι το τέλος ε, Δεκεμβρίου η, η συνολική αξία των Ε, συνολικών επενδύσεων των 12 ε, μεγαλύτερων ε, χωρών ανερχόταν σε σχεδόν 1 δισεκατομμύριο, 985 εκατομμύρια συγκεκριμένα. Το ΡΑΝ αυτή τη στιγμή, η ισοτιμία του ΡΑΝ με το ευρώ είναι 9,5. Έτσι λοιπόν έχετε μια ιδέα των ποσών. Η συμφωνία αυτή στόχο είχε την εξάλληψη εμποδίων στο εμπόριο, δηλαδή των δασμών μέσα σε ένα διάστημα 10 ετών ε, μέχρι το 2012 ε, τα προϊόντα της, ε, της Νοτιού θα απαλλάσσονται από δασμούς. Οι εξαγωγές έχουν διπλασιαστεί σχεδόν από 11 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ε, ευρώ το 2000 μέχρι 22 ε, εκατομμύρια το 2009 ως αποτέλεσμα της παγκοσμίου οικονομικής κρίσης και δημοσιονομικής κρίσης. Οι εισαγωγές και εξαγωγές για το διάστημα 2008-2009 έχουν πέσει. Ωστόσο τώρα βλέπουμε αντιστροφή της τάσης αυτής. Οι σημαντικότερες εξαγωγές της Νοτιού Αφρικής ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και γεωργικά προϊόντα, φάρμακα, ε, σίδηρος και χάλιβας, ε, ενώ οι εισαγωγές μας συμπεριλαμβάνουν μηχανήματα, οχήματα, συσκευές, υφάσματα, καύσιμα, επιστημονικά όργανα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην διαδικασία παραγωγής. Η συμφωνία της EDA ε, έχει συμβάλει στην εμβάθυνση των ε, σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νοτιού Αφρικής. Ε, υπάρχουν όμως παρόλα αυτά δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και θα το διαπιστώσετε και εσείς όσον αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εξαγωγείς της Νοτιού Αφρικής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αναφέρονται σε μελέτη για τις επιπτώσεις του TDCA. Κάποιες από αυτές είναι θέματα ε, διαπίστευσης ε, ε, έχουν επίσης να κάνουν με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα το μέτρο που απαιτεί την περιγραφή της χρήσης των παραστοχτών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων. Οι πολύπλοκες απαιτήσει Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, είναι δυσνόητες. Ε, υπάρχει ένα σύστημα ε, θα, θα, θέλαμε ένα σύστημα έγκαιρον, έγκαιρης προειδοποίησης για τις αλλαγές που θα ε, θεσπίζονται εντό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα πολύ σύντομα τώρα να αναφερθώ στις διαπραγματεύσεις ε, για την... για την προστασία των διανοητικών δικαιωμάτων. Ε, θα ξέρετε ότι εμείς συμμετείχαμε στην ΕΠΑ από την αρχή, ε, αλλά δεν υπήρχε νομική δέσμευση της Νοτιού Αφρικής να συμμετέχει στην ε, διαδικασία. Προσκληθήκαμε όμως ως παρατηρητές. Το 2006 οι υπουργοί οι ζήτησαν η Νότια Αφρική να γίνει πλήρες μέλος της ομάδας αυτής και να μην απλά παρατηρητής η Νότια Αφρική συμφώνησε διότι αυτό συνέπεσε με την ενδιάμεση αναθεώρηση του TDCA που απαιτούσε αναθεώρηση και του κεφαλαίου που είχε να κάνει με το εμπόριο. Έτσι λοιπόν γίναμε μέλος της διαδικασίας ε, EPA ε, για, την και, τις οικονομικές ε, συμφωνίες ε, και συμφωνίες εταιρική σχέσης. Το άρθρο 31 της συμφωνίας ΣΑΚΟ λέει ότι είναι υποχρεωτικό για όλα τα μέλη να διαπραγματεύονται ως ομάδα και όχι μεμονωμένα. Γι' αυτό η συμφωνία ΣΑΚΟΥ ζητάει μηχανισμό συνεννόησης μεταξύ των μελών. Φυσικά, όπως γνωρίζετε, οι διαπραγματεύσεις EPA ήταν προστατευμένες διαπραγματεύσεις, ε, όχι μόνο για την ομάδα αυτή, αλλά για όλες τις ομάδες ε, χωρών στην ε, Αφρικανική Ήπειρο. Ακόμα μας απασχολούν οι διαπραγματεύσεις αυτές. Θα γνωρίζετε ότι στη δική μας ομάδα πέρσι τον Ιούνιο τέσσερις από τις χώρες Τέσσερις χώρες υπέγραψαν την EPA, η Νότια Αφρική όμως ως μέλος της ΣΑΚΟΥ δεν υπέγραψε τη συμφωνία αυτή για διάφορους λόγους, ε, κυρίως επειδή υπήρχαν ακόμα κάποια εκρεμή ζητήματα στις διαπραγματεύσεις που έπρεπε να αντιμετωπιστούν προτού να μπορέσουμε να υπογράψουμε τη συμφωνία. Η υπογραφή της συμφωνίας όμως όσον αφορά την απόφαση την Ποτσουάνα, ε, Λεσόθο και Σουαζιλάνδη να υπογράψουν την ε, συμφωνία. Ε, η υπογραφή αυτή στόχο είχε να διασκεδάσει τις άλλων χωρών σχετικά με τις συμφωνίες αυτές που θεωρείται ότι υποσκάπτουν τις περιφερειακές της διαδικασίας περιφερειακής ολοκλήρωσης ε, στην ΣΑΚΟ. Ωστόσο, η Επίτροπος ε, Κάθριν Άστον ε, έγινε Επίτροπος Εμπορίου και προσπάθησε να σπάσει το αδιέξοδο, επισκέφθηκε την Νότια Αφρική και συναντήθηκε με υπουργού πέρσι το Φεβρουάριο, συμφώνησε να εξετάσουμε αυτά που θεωρούσε εκείνη άλλη τα θέματα στις διαπραγματεύσεις. Κατόπιν, στην Αμήβια είχαμε μια διαπραγματευτική σύνοδο και καταλήξαμε σε συμφωνία σε πέντε σημαντικούς τομείς όπου δεν μπορούσαμε να βρούμε συμφωνία νωρίτερα. Αυτά συμπεριλάμβαναν ε, εξαγωγικούς δεσμούς, ε, ασφάλεια των τροφίμων, ε, περιορισμούς στον όγκο και την ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων. Ε, το, η βασική κρεμότητα αυτή τη στιγμή είναι ο ορισμός ε, των συμβαλωμένων και οι ε, ρήτρε γεωργικών εγγύσεων. Στην επιστολή του 2009 η Επίτροπος Άστον ενημέρωσε τους Υπουργούς ότι μετά τις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν έτοιμη να προχωρήσει σε υπογραφή της ΕΠΑ. προσφέροντας ε, στην, ε, ίσους όρους με αυτούς που προσέφερε στην Ποσφάνα, Λισόθο, Μοζαμβίγη και Σουαζιλάνδη. Όσον αφορά τις ανησυχίες ε, της Ναμίμπιας και της Νότιας Αφρικής, είπε ότι και για τις χώρες αυτές θα προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις για την ΕΠΑ. Η Αγγόλα, Ναμίμπια και Νότια Αφρική ε, συμφωνήσαμε ότι οι νέες διατάξεις στους πέντε βασικούς τομείς που συμφωνήσαμε θα ενσωματωθούν στην αναθεωρημένη ΕΠΑ προτού να υπογραφεί το τελικό έγγραφο. Ωστόσο, μετά την ε, συνάντηση αυτή ε, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ε, οπισθοχώρησε και είπε ότι δεν μπορεί να αλλάξει τον όρο EPA. Αλλά είπε ότι οι νέες διατάξεις θα συμπεριληφθούν στο τελικό κείμενο. Παρότι η κοινή διακήρυξη επρόκειτο να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων, τελικά συντάχθηκε μονομερός από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό ε, δεν μας παρέχει καμία νομική ασφάλεια για να αποφύγουμε τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν ε, από την εφαρμογή της ενδιάμεσης ε, EPA αποφασίστηκε η εφαρμογή επικύρωση και κοινοποίηση των ΠΟΕ της ενδιάμεσης EPA να ανασταλεί. Η θέση αυτή ε, μεταφέρθηκε από τους Υπουργούς ε, Σάκου στον Επίτροπο Ντεχούχτ. Και είπαμε ότι η εφαρμογή της ενδιάμεσης ε, EPA θα οδηγούσαν σε διάσπαση της ΣΑΚΟΥ. Οι ενδοπεριφερειακές σχέσεις θα κατακαιρματιζόντουσαν αντί να ενισχυθούν, που ήταν ένας από τους βασικούς στόχους της EPA και τα θεσμικά μας όργανα ε, μπορεί να μην μπορούσαν να ε, αντισταθούν στις πιέσεις ε, που θα επέφερε η εφαρμογή της EPA. Ωστόσο, ο Επίτροπος Δεχούχτη είπε ότι στόχος Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η υπογραφή και εφαρμογή της ενδιάμεσης EPA. Μάλιστα, η απάντηση αυτή δεν απαντάει σε κανένα από τα ζητήματα που μας απασχολούν. Υπήρχε συμφωνία του 2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που ε, έδινε εντολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ευέλικτη στις διαπραγματεύσεις, αλλά η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελικά ήταν διαφορετική. Πριν από έξι εβδομάδες ή κάτι τέτοιο, μαζί με τους βουλευτές μας συζητήσαμε το θέμα αυτό στην Νότια Αφρική και Ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Νότια Αφρική έστειλε επιστολή στον ε, Επίτροπο Δεχούχτε ζητώντας να γίνει ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στους, ε, στον Επίτροπο Δεχούχτε και στους ε, υπουργούς ΣΑΚΟΥ EPA. Ως ομάδα EPA πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αναστείλουμε την εφαρμογή και την επικύρωση και να έχουμε ε, τον χρόνο να εξετάσουμε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που εκκρεμούν. Μετά από διάστημα 14 μήνο, δεν βλέπουμε να υπάρχει καμία κίνηση. Οι αξιωματούχοι μας συναντήθηκαν το προηγούμενο μήνα Ελπίζουμε ότι με καλή βούληση από όλε τι πλευρέ θα μπορέσουμε να κινήσουμε τη διαδικασία και σε σύντομο χρονικό διάστημα να μπορέσουμε να λύσουμε τις εκκρεμότητες και να έχουμε μια πλήρη EPA που να καλύπτει προϊόντα, και αγαθά και υπηρεσίες μέσα σε λογικό χρονικό διάστημα. Θα κλείσω εδώ. Ε, έχω εδώ μαζί μου το που είναι επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικού Εμπορίου. Έχουμε την... Έχω και τις δύο συνεργάτητές μου που συμμετέχουν στην διαδικασία EPA. Σας ευχαριστούμε και πάλι που μας δώσατε την ευκαιρία να παρευρεθούμε εδώ. Well, let's open the uh, exchange of views. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με την ανταλλαγή απόψεων. Ξεκινάμε με τα μέλη της Επιτροπής μας. Η κυρία Μουσκαρντίνη από το ΕΛΚ καταρχάς. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Πρέσβη για την πολύ συγκεκριμένη αυτή παρουσίαση που κάνατε, την οποία νομίζω ότι θα πρέπει να μελετήσουμε πολύ προσεκτικά, ιδίως τα όσα μας είπατε για την Συμφωνία Οικονομικής οικονομικής-στερικής Σχέσης, αλλά και για το ΣΑΚΟΥ, την Τελωνιακή Ένωση της Νότιας Αφρικής είναι ζητήματα τα οποία μας απασχολούν πάρα πολύ. Και ουσιαστικά τα όσα είπατε έχουν να κάνουν με το ρόλο που θέλει να διαδραματίσει η Νότια Αφρική προκειμένου να καταφέρει να καταλήξει σε μια επιτυχή εξέλιξη του διαπραγματευτικού γύρου της Ντόχα. Στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία είχα παρακολουθήσει πάρα πολλές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια της Επιτροπής αυτής και είχαμε πάρα πολύ τη δυνατότητα να εξετάσουμε για παράδειγμα μια πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις απαραίτητες τροποποιήσεις που έπρεπε να γίνουν στο διεθνές εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου η Νότια Αφρική να μπορεί να συμφωνεί με τη στάση που ήθελε να προωθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή να μην μπαίνουν όλες οι χώρες ε, στο ίδιο επίπεδο, δηλαδή να γίνει ένα διαχωρισμό ανάμεσα στι χώρε εκείνε που παρουσιάζουν πλέον μια έντονη οικονομική ανάπτυξη και τι χώρε εκείνε οι οποίε υστερούν οικονομικά. Θα ήθελα να γνωρίζω επίση και την άποψή σα για τον κύκλο διαπραγματεύσεων τη Ντόχα. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο συζητήσαμε και με τον Επίτροπο Ντεγκούχτ είναι ότι στην Αφρικανική Ήπειρο το τελευταίο καιρό δύο πολύ οικονομικά ισχυρές χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία ξεκίνησαν μία πολιτική θα έλεγα ιδιαίτερα επιθετική ή τουλάχιστον πολύ ισχυρή αν θέλετε στην εξαγορά γέας, αλλά, γεών, με συγχωρείτε, αλλά και στις εμπορικές ανταλλαγές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικός εταίρος της ε, Αφρικανικής Υπήρου και συγκεκριμένα της Νοτιού Αφρικής Θέλουμε να έχουμε πάντα πιο εδρεωμένες και ισχυρές σχέσεις μαζί σας. Θα θέλαμε όμως να γνωρίζουμε και τη δική σας άποψη όσον αφορά την επιθετική αυτή προσέγγιση της Ινδίας και της Κίνας. Επιθετική σε σχέση και με τη δική μας προσέγγιση, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή. Και πώς αυτό θα δημορφώσει το οικονομικό μέλλον της συνεργασίας μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά την EPA, πιστεύω ότι θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να υπογράψουμε η EPA με όσο γίνεται περισσότερες χώρες και να μην μείνουμε στις ενδιάμεσες EPA. Διότι στον τελωνιακό χώρο της ε, κοινότητας για την ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής ε, βλέπουμε την τάση να υπογράφονται συμφωνίες με κάποιες χώρες και με άλλες όχι. Κύριε Πρόεδρε, θα θέλαμε όσο γίνεται πιο γρήγορα να έχουμε τη δυνατότητα να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να συζητήσουμε μια οριστική EPA με την παράδοση που έχουμε στις διαπραγματεύσεις μας με την Νότια Αφρική. Πιστεύω ότι έχει δημιουργηθεί εμπιστοσύνη και ότι έχουμε επιφέρει έτσι πολλές θετικές οικονομικές αλλαγές στην Νότια Αφρική. Οι διαπραγματεύσεις κατά τη δεκαετία του 1990 δεν ήταν απλές. Τέσσερα χρόνια διήρκησε η επίτευξη συμφωνίας με την Νότια Αφρική. Ωστόσο, Δεν θα πρέπει να διακυβεύσουμε την κατάσταση με την προώθηση των ενδιάμεσων EPA, ε, αφήνοντας έξω άλλες ενδιαφερόμενες χώρες. Μία ερώτηση έχω για ένα άλλο θέμα. Η ζάχαρη μέχρι τώρα δεν έχει ενσωματωθεί στην εμπορική συμφωνία. Έχω λάβει πληροφορίες από την Νότια Αφρική ότι οι μικροί γεωργοί ε, συμμετέχουν στην ε, παραγωγή ζάχαρης λόγω της, μεταρρυθ... λόγω γεωργικής μεταρρύθμισης και ότι η συμπερίληψη της ε, ζάχαρης στη... στο εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενίσχυε την θετική αυτή εξέλιξη. Μήπως μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε πρέσβη. Οργανώσετε ένα παγκόσμιο κύπελο ράγμπι και ένα παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και τις δύο φορές ιτήθηκε η Γαλλία. Λοιπόν, πολιτικά είναι πολύ ισχυρό το θέμα. Εγώ υποστήριξα την Νότιο Αφρική κατά της Γαλλίας για το ποδόσφαιρο, αλλά κοιτάστε, δεν πρέπει να γίνει συνήθεια αυτή η στάση. Επί της ουσίας. Η Νότια Αφρική στα πλαίσια των εμπορικών συναλλαγών της ΠΟΕ ε, είναι τμήμα αυτών των χωρών που επέμειναν πάρα πολύ στην ε, μεγάλη απολευθέρωση στον τομέα της γεωργίας. Εμείς σήμερα από την ευρωπαϊκή πλευρά ακούμε ότι για να βγούμε από το διέξοδο των διαπραγματεύσεων στην ΠΟΕ θα πρέπει να βγούμε από αυτήν την περιορισμένη ατζέντα για τις ε, υπηρεσίες και περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Θέλω να ξέρω αν η προπτική μιας περιορισμένης ημερήσιας διάταξης είναι κάτι το οποίο το έχει κατά νου ή είναι αποδεκτό τέλο πάντων για την ε, Νότια Αφρική. Η Νότια Αφρική μαζί με την Κίνα, την Ινδία, την Βραζιλία βαραίνουν ιδιαίτερα στον ορισμό για το τι μπορεί να αποτελεί σήμερα την πολυμερότητα. Εμείς το είδαμε στις διαπραγματεύσεις ε, στην Κοπενχάγη η Κίνα συμμετείχε ίσως μαζί με τις Ηνωμένε Πολιτείες σε μια άλλη οπτική για την πολυμερότητα, δηλαδή ένα gentleman agreement, μια συμφωνία κυρίων σε διεθνές επίπεδο, και είχαν ένα όραμα όπου τα κράτη-μέλη δεσμεύονται ατομικά και το διεθνές πλαίσιο θα αποτελούσε ε, το χώρο ε, καταμερισμού αυτών των ε, ε, ατομικών επιλογών και ανακοίνωσης των, κοινών επιλογών και όχι την αποδοχή μιας κοινή ευθύνης που αναλαμβάνουμε όλοι και την εφαρμόζουμε όλοι. Ποια είναι η θέση της Νότιας Αφρικής σχετικά. Επίσης η Ευρώπη χρησιμοποιεί, θεσπίζει σήμερα κριτήρια ας πούμε για τα βιοκάψιμα ε, δηλαδή την αηφορία τη θεωρεί κριτήριο για τις, ε, για τις διμερείς συμφωνίες. Εσείς θεωρείτε ότι θα μπορούσατε να το δεχτείτε. Σας ευχαριστούμε. Θα πρέπει να δώσουμε και τον απαραίτητο χρόνο στον πρέσβη να απαντήσει στις ερωτήσεις. Επομένως, οι υπόλοιποι ομιλητές πρέπει να μιλήσουν πολύ σύντομα. Σας παρακαλώ, κύριο Κάμπελ. Κύριε πρέσβη, θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο σημαντικό είναι ε, για το εμπόριο της Νοτιής Αφρικής η θέση που έχετε εσείς στην κοινοπολιτεία. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε καταρχάς βέβαια στην Ινδία, η οποία το 2050 θα έχει γίνει η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίω. Οι δικέ σα εμπορικές πρακτικές, η δική σα η γλώσσα, η νοοτροπία που υπάρχει στην Νότια Αφρική μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό πλεονέκτημα στα πλαίσια τη κοινοπολιτεία. Ο κύριος Ράμστον, σας ε, ευχαριστώ. Ε, αναφερόμαστε κοινοπολιτεία, αλλά τελικά δεν υπάρχει κοινό παράγοντα στα πλαίσια του εμπορίου στην κοινοπολιτεία. Θα ήθελα να συγχαρώ τον ε, πρέσβη της Νοτιού Αφρικής και γενικά τους ηθήνοντες στην Νότια Αφρική για την διοργάνωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου μπορεί να έχουν ε, διανύσει ε, δύσκολες ε, εποχές, αλλά το σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι την εποχή της ανοικοδόμησης και της αναδιάρθρωσης στη χώρα γνώρισαν και πολλά δημοσιονομικά προβλήματα. Ο Τζένεραν Μάλιον κατάφερε να διατηρήσει την σταθερότητα στην Νότια Αφρική, στο νοτιοαφρικανικό κράτος και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Το ερώτημά μου είναι το ακόλουθο. Πώς μπορούμε να διατηρήσουμε την μακροοικονομική σταθερότητα της Νοτιοαφρικής προκειμένου να πραγματοποιήσει τα φιλόδοξα προγράμματά της για την ανοικοδόμηση και την διάρθρωση στις ε, υφιστάμενες περιστάσεις και το άλλο ζήτημα στο οποίο θα θέλω να θίξω είναι η μεταναστευτική πίεση. Η Νότιος Αφρική αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα στην ολοκλήρωση και την ανάπτυξη της Αφρικανικής Υπήρου εν γέννη. Η Νότιος Αφρική όμως είναι και μια χώρα που εκτίθεται σε πολύ έντονες μετνευστικές πιέσεις από όμορες χώρες και τον Μάιο του 2008 γίναμε μάρτυρες διενέξεων, συγκρούσεων ανάμεσα σε ηθήνοντες της Νοτιοαφρικής και μετανάστες κυρίως από την Τζιμπάμπουε. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις αρνητικές επιπτώσεις από την μετνεστευτική πίεση. Ο κύριος ε, Στανσνή από το ΕΛΚΑ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε, σας ε, ευχαριστώ κύριε πρέσβη. Θα ήθελα και εγώ όπως και προλύσαντες να σας ε, συγχαρώ για την καταπληκτική διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Όλοι όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε πρόκειται για εφημερίδες, είτε πρόκειται για ραδιόφωνα τηλεοράσεις, είπανε ότι η διοργάνωση ήταν καταπληκτική. Ελπίζω να καταφέρετε να πάρετε και του Ολυμπιακού του 2020. Ξέρω ότι ε, ε, φέλησε πάρα πολύ την Νότιο Κορέα, φέλησε πάρα πολύ το Σίδνεϊ και γενικά όλες τις πόλεις οι οποίες κατάφεραν να κερδίσουν τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Σας εύχομαι λοιπόν και σε εσά να μπορείτε να υποδεχθείτε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020. Έχετε φτάσει πλέον στο επίπεδο των ε, ηγετικών κρατών σε παγκόσμιο επίπεδο. Δείχνετε μια ηγετική θέση, διαδραματίζετε έναν ηγετικό ρόλο. Αυτό περιμένει η εταίροι σας, αυτό περιμένουν από εσά οι υπόλοιπε χώρες και καταφέρνετε να δεξάγετε το ρόλο αυτό πάρα πολύ καλά. Επομένως απευθύνονται σε εσά ρωτώντας σας ε, τι μπορεί να γίνει στα πλαίσια της ε, συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι η συμφωνία αυτή, το είπατε και ο ίδιος, για τη γενικότερη περιφέρεια της Μεσημβρινής Αφρικής. Είναι όμως και μια συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μπορεί να ωφελήσει όλη την Αφρικανική Ήπειρο. Σε εσά ουσιαστικά απευθύνονται οι εμπορικοί σας εταίροι στην Αφρική προκειμένου να καταφέρετε να αναβαθμίσετε όλη την Ήπειρο. Στην πράξη όμως, πώς καταφέρνετε να καταπολεμήσετε τη διαφθορά. Η διαφθορά είναι βέβαια ένα παγκόσμιο πρόβλημα, αλλά εντοπίζεται ιδιαίτερα στην Αφρικανική Ήπειρο. Όταν είδα για παράδειγμα την υπερτιμολόγηση που γίνεται για διάφορα έργα υποδομής στην Αφρική που φτάνουν πολλές φορές και τα δισεκατομμύρια, αναρωτήθηκα ακριβώς αυτό το πράγμα τι μπορεί να κάνετε εσείς για τα δύο αυτά ζητήματα, την καταπολέμηση τη διαφθοράς και τον ηγετικό ρόλο που δείχνετε στα πλαίσια της ΕΠΑ, τη Συμφωνίας Οικονομικής εταιρική σχέση. Σας ευχαριστώ. I, I will be very brief. Θα είμαι πολύ σύντομο ε, κύριε Πρόεδρε. Ζητώ... Φοβάμαι... Λυπάμαι που θα είμαι ο πρώτος ε, με τα άσχημα νέα, διότι αμφισβητώ το ποσό των χρημάτων που ε, δαπανήθηκε για τη διοργάνωση του ε, παγκοσμίου κυπέλου, διότι είδαμε νέα στάδια και ένα σωρό υποδομές, ενώ πάρα πολλοί νοτιοαφρικανοί δεν έχουν ε, στέγη πάνω από το κεφάλι τους. Κατά τη γνώμη μου αυτό δεν είναι λόγος για συγχαρητήρια. Κάποιοι κέρδισαν πολλά από αυτό, αλλά ε, οι περισσότεροι Νοτιοαφρικανοί όχι. Εμένα με ενόχλησε επίσης πάρα πολύ ότι υπήρξε ποινικοποίηση ε, τα θεμητών και ειρηνικών διαδηλώσεων. Προδίδεται όλες τις παραδόσεις της εργατικής τάξης της ε, Νοτιού Αφρικής και τους αγώνες που ε, έκανε κατά, της, ε, κατά τους καθεστώτος Apartheid. Κύριε Πρέσβη, μπορείτε να είσαστε πιο συγκεκριμένοι όσον αφορά τα εκρεμή ζητήματα που αναφέρατε επανειλημμένα όσον αφορά τις δυσκολίες της Νοτιού Αφρικής με τη Συμφωνία EPA. Ποια ακριβώς είναι τα ζητήματα αυτά, μπορείτε να είστε πιο συγκεκριμένος και όσον αφορά τις χώρες που είναι έτοιμε να υπογράψουν το EPA, ποια είναι η σχέση σας με αυτές για τα ζητήματα αυτά και άλλα ζητήματα. Τέλος, Στι ε, μελλοντικέ εμπορικέ σχέσεις θα ήθελα να σα ρωτήσω ποια είναι η θεμελιώδης φιλοσοφία της ε, κυβέρνησης της Νοτιού Αφρικής. Το, ε, ε, το ANC ήταν ε, προοδευτικό αριστερό ε, κόμμα όσον αφορά την οικονομική πολιτική. Ποια είναι η θέση τώρα της κυβέρνησης απέναντι στην ε, ιδιωτικοποίηση, απελευθέρωση των ε, υπηρεσιών κλπ. και στα πλαίσια των εμπορικών συμφωνιών και πώς ε, ωφελεί αυτό τα εκατομμύρια φτωχών στην Νότια Αφρική. Ευχαριστώ πολύ. Για να κλείσουμε τη συζήτηση, θα, δώσω το, για να κλείσουμε τον κύκλο αυτό, θα δώσω το λόγο στον Μάικλ Κάσμαν, που συμμετέχει στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σχέση με την ε, Νότια Αφρική. Καθότι ήδη έχουμε καθυστερήσει, σας παρακαλούσα να είστε σύντομος. Νομίζω ότι θα αποδείξω ότι πράγματι ε, ε, ούκαν το πολλό το ΕΦ. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε στην συνεδρίασή σας. Θα ήθελα να αναφερθώ στα, στις συμφωνίες EPA. Πρόσφατα επισκεφθήκαμε την Νότια Αφρική και πρέπει να πω ότι οι επενδύσεις στην υποδομή φαίνεται να ωφελούν και άλλους πέρα από τους, ε, αυτούς που έκαναν τα έργα και φαίνεται να το βλέπουν θετικά οι πολίτες της ε, Νοτιού Αφρικής. 25 ε, και 26 Μαΐου είχαμε συζητήσεις με τους βουλευτές και οι δύο πλευρές έδειξαν το θέμα των συμφωνιών EPA. Στείλαμε επιστολή στον Καρλ Ντεκούχτ, ε, λέγοντας ότι πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει η υπουργική συνάντηση υψηλού επίπεδου ανάμεσα σε αυτόν και στους ε, υπουργού ΣΑΝΤΑ και EPA για να ε, εκφραστεί η πολιτική βούληση για επιτυχή ολοκλήρωση. Χαίρομαι που είχαμε θετική απάντηση και να σας πω τα βασικά. Ο Επίτροπος προσλέπει στην μελλοντική διάσκεψη κορυφής ευρωπαϊκή Ένωσης Νοτιού Αφρικής ως ευκαιρία για να αξιολογήσει την ε, κατάσταση και επίσης ε, ε, εξερευνά τη δυνατότητα να υπάρξει συνάντηση με τις χώρες σαν και EPA μετά το καλοκαίρι. Είναι λοιπόν πολύ θετικέ οι εξελίξεις. Επικροτώ την επίσκεψη της Επιτροπής σας το ταξίδι που οργανώνει η Επιτροπή σας. Πιστεύω ότι έτσι θα ενισχυθούν οι προσωπικές και πολιτικές σχέσεις που έχουμε δημιουργήσει και πιστεύω επίσης ότι θα οικοδομείται στην ειλικρίνεια με την οποία η κάθε πλευρά αντιμετωπίζει τα προβλήματα ώστε να συμμετέχουμε όλοι στην εξέβρεση λύσης. Επίσης θα σας παρακαλούσα να με ενημερώσετε σχετικά με την επίσκεψή σας. Νομίζω ότι είναι προαιρετική δική μου συμμετοχή αλλά πιο σημαντικό είναι το ότι αν με ενημερώσετε, πολύ ευχαρίστω θα σας βοηθήσω με οποιονδήποτε τρόπο μπορώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρέσβη για τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο πάντα είχε επαφές με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Μάικλ. Πάντα χαιρόμαστε να ακούσουμε τις παρεμβάσεις σας να δώσω τώρα το λόγο στον προσκεκλημένο μας ε, για να απαντήσει στις πολλές ερωτήσεις και παρατηρήσεις που του απευθύναμε. Είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσετε να απαντήσετε μέσα σε ένα λογικό χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω για δύο λεπτά και μετά θα δώσω το λόγο στον συναδελφό μου. Πολύ σύντομα να πω ότι όσον αφορά το ρόλο της Νοτιού Αφρικής στην Ήπειρο αυτή, όταν γίναμε δημοκρατία, δεν επικεντρωθήκαμε αποκλειστικά σε εσωτερικά ζητήματα. Αναγνωρίσαμε ότι έχουμε να παίξουμε πιο σημαντικό ρόλο, όσο και αν μας τύχει αυτό. Ναι, έχουμε φτώχεια, ε, υποανάπτυξη στη χώρα μας. Ε, αυτό το βλέπει η παγκόσμια κοινότητα, δεν το κρύψαμε ποτέ. Αντιμετωπίζουμε τεράστιες προκλήσεις, πολλές από τι οποίε τι κληρονομήσαμε. Ενώ άλλες ε, δημιουργήθηκαν ε, κατά την ανάπτυξή μα. Δεν πιστεύουμε σε μια μονομερή παγκόσμια κοινότητα. κοινότητα. Η Νότια Αφρική πιστεύει στην πολυμερή παγκόσμια κοινότητα. Παρότι συμμετέχουμε σε κάποιες ε, ομάδες όπως η Κοπεχάγη, η Ήψα, ε, η Νότια Αφρική κλπ. Όλα αυτά γίνονται για να ενισχύσουν περαιτέρω την πολυμέρεια. Για μας αυτή η πολυμερής προσέγγιση είναι το κλειδί για την εξωτερική πολιτική. Και θα ήθελα επίσης να πω ότι η Νότια Αφρική παίζει ρόλο για την ειρήνη και σταθερότητα στην Ήπειρο. Καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε μία νησίδα πλούτου σε έναν ωκεανό φτώχεια γι' αυτό. Η δέσμευσή μας δεν είναι μόνο απέναντι στην Νότια Αφρική αλλά και στην περιφέρειά μας και στην η ε, πυρό στο σύνολό της. Δισεκατομμύρια ραν ξοδεύουμε, ε, χρήματα που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν, θα μπορούσε να πει κανεί για να αντιμετωπίσουμε ε, εσωτερικά προβλήματα. αλλά ξοδεύουμε πολλά χρήματα και σε άλλα μέρη της Υπήρου, στην Ζιμπά, που ε, ή Το θέμα είναι λοιπόν ε, πού θα επενδύσει κανείς τους πόρους του. Ε, θα έχουμε εσωστρεφή οπτική, θα χτίσουμε για μας υποδομή, στάδια κλπ και θα επικεντρωθούμε στις ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην πατρίδα μας. Ε, δεν είναι αυτή η πολιτική της Νοτιού Αφρικής. Ε, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα εσωτερικά μας προβλήματα αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι είμαστε μέλος της Υπήρου της Αφρικής και ότι τα προβλήματα της Αφρικής είναι και προβλήματα της Νοτιού Αφρικής. Η Αφρική θα πρέπει να γίνει αναγνωρισμένο μέλος της ε, παγκόσμιας κοινότητας ε, και στο εμπόριο και στο, στην πολιτική και στον αθλητισμό. Αυτό κινεί την Νότια Αφρική. Όσον αφορά τον ε, γύρο της Δόχα, θα ζητήσω από τον συνάδελφο να πάρει το λόγο. Η δέσμευσή μας υπάρχει. Πάντα παίζαμε σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ. Είναι αναπτυξιακός γύρος και θέλουμε να ε, συμβάλλουμε σε αυτό. Ε, επειδή δεν έχουμε χρόνο θα κλείσω εδώ και θα ζητήσω από τον συνάδελφό μου να πάρει το λόγο. Όσον αφορά τον κύκλο διαπραγματεύσεων της ΔΟΧΑ θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η Νότιος Αφρική υποστηρίζει αυτόν τον κύκλο διαπραγματεύσεων και συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να καταλήξουμε γρήγορα σε μια θετική έκβαση σε αυτόν τον γύρο διαπραγματεύσεων. Πραγματικά πιστεύουμε ακόμα ότι μπορούμε να καλύψουμε όλες τις πτυχές διαπραγματεύσεων δεν υπάρχει λόγο σε αυτή τη φάση τουλάχιστον να περιορίσουμε τι προτεραιότητέ μα και την ατζέντα. Στόχο είναι να ανταποκριθούμε στι ανάγκε των αναπτυσσομένων κρατών και όπω είπε και ο πρέσβη μα, στόχος μας είναι οι πολυμερείς εμπορικές σχέσεις οι διμερείς εμπορικές σχέσεις είναι δευτερεύουσα σημασία για μα. Αυτό το οποίο θέλουμε εμεί να προωθήσουμε και αυτό που τελεί για μα προτεραιότητα είναι οι πολυμερει εμπορικές συμφωνίες σε επίπεδο παγκόσμιου οργανισμού εμπορίου. Προσπαθούμε σε διμερές επίπεδο να έχουμε περιορισμένη ατζέντα γιατί δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει λόγο να έχουμε σε παγκόσμιο επίπεδο μια πληθώρα διμερών εμπορικών συμφωνιών. Ένα βουλευτή αναφέρθηκε στο ζήτημα της ζάχαρης. Όπως γνωρίζετε, η Νότιο Αφρική αποτελεί θύμα αρνητικής διακριτικής μεταχείρισης σε σχέση με άλλε συναπτυσσόμενε χώρε οι οποίε στι εμπορικέ συναλλαγέ που έχουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν προνομιούχο θέση όσον αφορά το ζήτημα τη ζάχαρη και τι εξαγωγέ που κάνουν σε ζάχαρη από τι χώρε αυτέ προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια της μεταρρύθμισης που έλαβε πρόσφατα χώρα στη Νότια Αφρική όσον αφορά την γεωργία μας και την χωροταξία, θελήσαμε να προωθήσουμε και τα δικά μας προϊόντα ζάχαρης και να έχουμε ισότιμη πρόσβαση με τις άλλες χώρες. Όσον αφορά τα ζητήματα που δεν έχουν επιληθεί στην EPA, είναι καταρχάς η πρόσβαση στις αγορές, η Νότιος Αφρική κατά τη διαπραγμάτευση τη Συμφωνίας για το Εμπόριο, την Ανάπτυξη και τη Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε περιορισμένη πρόσβαση στη φάση εκείνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως όσον αφορά στις ε, αγορές γεωργικών προϊόντων. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα επιληθεί το πρόβλημα αυτό και ότι όπως μας είχατε υποσχεθεί τότε θα ανοίξετε περισσότερο την πρόσβαση στα δικά μας προϊόντα. Επίσης περιορίζεται η σχέση εμπορικών συναλλαγών που έχουμε με τρίτες χώρες στα πλαίσια της EPA και ένα τρίτο ζήτημα που δεν έχει επιληθεί είναι η νέε δομέ με τι οποίε εμεί θα πρέπει να ευθυγραμμιστούμε, είτε ότι μα ζητάτε να δημιουργήσουμε νέου θεσμού. Εμεί ήδη έχουμε τη ΣΑΚΟΥ, την Τελωνιακή Ένωση Νότια Αφρική, καθώ επίση και την SADC, την Κοινότητα για την Ανάπτυξη τη Μεφρεσνή Αφρική. Λειτουργούν πολύ καλά οι θεσμοί αυτοί. Δεν υπάρχει λόγο να δημιουργήσουμε νέου. Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη, σα ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ και τους συνεργάτες σας που ήρθαν στη συνεδρίαση. Προφανώς αυτή την είναι η τελευταία επαφή που θα έχουμε. Θα μείνουμε σε επαφή, θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας, θα προετοιμάσουμε μαζί και τις συνεδριάσεις της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νοτιοαφρικής. Πρόκειται για την πρώτη αποστολή, την πρώτη προσωπία που θα έχουμε στην Νότια Αφρική, αυτή την οποία προετοιμάζουμε. Επομένω, θα ήθελα πραγματικά να στεφθεί με επιτυχία και βασιζόμαστε και στη δική σα τη συμβολή προκειμένου να επιτύχει να είναι επικοδομητική επίσκεψη που θα πραγματοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται κατά αυτόν τον τρόπο η συνεδρίασή μας. Βέβαια έχουμε ένα ακόμα σημείο το οποίο θα καλυφθεί και κλεισμένο το θυρών. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Ντέιβιτ Οσάλιβαν, το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου της Επιτροπής. Θα ήθελα σε όσους θα αποχωρήσουν να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές. Παρακαλώ πολύ, απαχωρήστε από την αίθουσα όσο το δυνατόν συντομότερα. Και όλες αυτές οι συζητήσεις να γίνουν εκτός αιθούσας, παρακαλώ.